Καλημέρα, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ακόμα δεν έχουν έρθει όλοι για να κάνουμε την πλήρη συζήτηση. Είναι πρώτη και τελευταία φορά που έχουμε παράλληλη συνεδρίαση με την Επιτροπή Προϋπολογισμών αλλά πολλοί συνάδελφοι εδώ στην Επιτροπή δεν είναι μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμού και για αυτούς δεν υπάρχει δικαιολογία. Πρέπει να αρχίσουμε στην ώρα μας γιατί ο εισηγητής θα είναι στη διάθεσή μας μέχρι τις 11 και μετά δυστυχώς πρέπει να φύγει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις μας και θα κρίνουμε αν υπάρχουν κι άλλες ανάγκες ή αν μπορούμε να ολοκληρώσουμε εκείνη την ώρα τις συζητήσεις μας. Θα δούμε, είμαστε αρκετά ευέλικτοι και ταχύς. Αυτό διέκρινε πάντα την Επιτροπή ΣΟΥΡΕ. Μετά από αυτό έχω μία ανακοίνωση μόνο. Όλα τα άλλα θα τα κάνουμε μετά το τέλος αυτής της συζήτησης, ό,τι χρειάζεται να ανακοινωθεί δηλαδή. Και τώρα θα ήθελα να πω κάτι για την δομή της συζήτησής μας εδώ. Ξέρετε ότι έχουμε περίπου 1.100 τροπολογίες που δεν μπορούμε να τις συζητήσουμε σε μια συνεδρίαση όλες, ούτε μπορούμε να επισέλθουμε σε κάθε μία χωριστά. Πρέπει λοιπόν να δομήσουμε την συζήτηση σε τρία μέρη μάλιστα. Με βάση την ε, επιθυμία μας να διατηρήσουμε τη δομή της έκθεσης με τα έξι κεφάλαια και τους έξι τίτλους. Αυτά θα μείνουν ως έχουν και σε τρία μέρη θα χωρίσουμε τη συζήτηση για τις τροπολογίες. Ο εισηγητής προφανώς θα μας κάνει μια γενική εισαγωγή και θα κάνει και γενικά σχόλια. Μετά όμως θα πιάσουμε το πρώτο μέρος της έκθεσης για τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες Στην έκθεση αυτή, ε, το κομμάτι αυτό είναι μέρος 1 με 3. Μετά, στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, θα συζητήσουμε το τμήμα ή το μέρος 4 της έκθεσης για τη δομή, την οργάνωση και τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές και το μέρος 5 της έκθεσης θα το συζητήσουμε στο τρίτο μέρος της συζήτησης. Το αντικείμενο είναι να δούμε τη σχέση μεταξύ εσόδων και δαπανών για να δούμε την τάξη μεγέθους των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών και τους δικούς μας ίδιους πόρους. Κατόπιν τούτου θα παρακαλέσω τον εισηγητή να κάνει το γενικό εισαγωγικό μέρος, πέντε λεπτά κάθε φορά και μετά θα περνάμε στο γύρο της, ε, των παρεμβάσεων των ε, αγοριτών από τις πολιτικές ομάδες και κατά δεύτερο λόγο θα δώσουμε το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους. Σαλβαντόρ παρακαλώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ Πρόεδρε, ούτως ή άλλως είμαι ευέλικτο. Ε, ε, Όπως ελέγχθη θα ήθελα να φύγω στις 11, αλλά εν πάση περιπτώσει αν ε, χρειάζεται να μείνω επιτακτικά θα αλλάξω τα σχέδια μου και θα μπορέσω ίσως να μείνω περισσότερο ώστε να μπορέσουν όλοι οι συντονιστές και οι συνεισηγητές να παρουσιάσουν το θέμα. Θα ήθελα σε γενικές γραμμές να πω ότι η έκθεση της Επιτροπής ΣΟΥΡ είναι μια πολιτική δήλωση του Κοινοβουλίου για τις ε, μελλοντικές χρημα... οικονομικές προοπτικές. Πολλές φορές ανέφερα το γεγονός ότι θα πρέπει η ψηφοφορία να έχουμε γύρω στους 50 ψήφους. Δεν είμαι ματαιόδοξος, ούτε υπερόπτης. Απλώς θα πρόκειται για γενικότερη ε, συνένεση στο Ευρωκοινοβούλιο και θα μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να έχουμε πραγματικές σημαντικές επιπτώσεις και επιτροπής και για τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν για το πρόξιμο πολιετές πρόγραμμα που θα αρχίσουν το Συμβουλίο το Σεπτέμβριο. Έχουμε 1093 τροπολογίες περισσότερες δεν ε, εισαγάγουν ριζικές αλλαγές, απλώς πρόκειται για βελτιώσεις. Υπάρχουν ε, ώρες ώρες και κάποιες διθέσεις θέση μου και πιστεύω ότι για τα περισσότερα θέματα μπορούμε να καταλήξουμε σε συνένεση. Ο τρόπος με τον οποίο δούλεψαν οι πολιτικές ομάδες είναι πολύ χρήσιμος, διότι επιτεύχθηκε και στις ίδιες πολιτικές ομάδες εσωτερική συνένεση και έτσι ε, κατατέθηκαν στον εισηγητή εκ μέρους των πολιτικών ομάδες, ε, ομάδες ολόκληρα μπλοκ τροπολογιών. Έτσι μπόρεσα να κάνω μια πρώτη σειρά συμβαστικών τροπολογιών ώστε να απλοποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσω να συγκεράσω τις διάφορες πολιτικές απόψεις στην έκθεσή μου. Υπάρχουν κάποιες ε, τροπολογίες που κατέθεσαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν είναι μέλη της Επιτροπής ΣΟΥΡ, στις οποίες παρουσιάζονται λεπτομέρειες για τα διάφορα θέματα τα οποία μελετούμε εμείς. Πρόκειται όμως για πάρα πολύ μεγάλες λεπτομέρειες. Δεν είναι θέμα διαφορών σημαντικών, αλλά αν μπούμε σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες και τις αποδεχθούμε, νομίζω ότι θα μπούμε στα χωράφια κατά κάποιο τρόπο άλλων επιτροπών. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι είναι σωστό τρόπο. Σε πάση περιπτώσει, εγώ ότι αφορούσε τον προπολογισμό, πιστεύω ότι θα πρέπει να το εγκρίνουμε και όλες τις άλλες λεπτομέρειες, όπως είπα, να τις αφήσουμε στις αρμόσιες επιτροπές. Επίσης, ξέρουμε ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει 150 παραγράφους η έκθεση Διαφορετικά θα είναι αντιπαραγωγικό το έργο που κάνουμε. Ξέρουμε ότι κατατέθηκαν πάρα πολλές τροπολογίες ε, από τις πολιτικές ομάδες και από τα μέλη της Επιτροπής σουρε αλλά ελπίζω ότι θα είμαστε αρκετά ευέλικτοι όλοι για να μπορέσω εγώ να κρατήσω αυτή την δομή της εκθεσή μου και κατά το τώρα της 150 παραγράφους. Όπως είπε και η Πρόεδρος, επίσης θα ήθελα να διατηρήσω παρούσα δομή της ε, έκθεσης. Έχει την ενοποιημένη παρουσίαση της έκθεσης αναλάβει η γραμματεία, ώστε να είμαστε και συνεκτικοί με το, με το πιστοτικό ε, πλαίσιο. Όπως σας είπα, θα παρουσιάσω πολλές τροπολογίες ε, συμβιβαστικές για να μπορέσουν να αντικατοπτριστούν όλες οι απόψεις των πολιτικών ομάδων. Κάναμε μια πρώτη αξιολόγηση των τροπολογιών στις πολιτικές ομάδες και όσον είδαμε, για τα περισσότερα θέματα υπάρχει μεγάλη σύγκληση μεταξύ των μεν και των δε. Βεβαίως, για κάποια θέματα δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στη συνένεση, άρα θα πρέπει να κάνουμε πιο ενδελεχή συζήτηση για αυτές, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα κύρια θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και θα υποβάλουμε σε ψηφοφορία. Στις 24 ε, και 25 Μαΐου στη συνεδρίασή μας θα πρέπει να έχουμε τις λιγότερες δυνατές τροπολογίες και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις παρατηρήσεις, στις ανησυχίες που εξέφρασαν οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ. Ο συντονιστής του ΕΛΚ δεν είναι εδώ. Θα αρχίσουμε με τον συντονιστή των ε, σοσιαλιστών κατά πρώτο λόγο λοιπόν. Δεν είμαστε έτοιμοι για τη συζήτηση αυτή. Θεωρούσαμε ότι θα γίνει η συζήτηση τώρα για τις προκλήσεις και τις πολιτικές προτεραιότητες. Ήρθε η ώρα τώρα ή όχι ακόμα. Όχι, τώρα θα κάνουμε γενικά σχόλια. Καλά, θα κάνω λοιπόν γενικά σχόλια και θα συνεχίσουμε μετά. Γενικό σχόλιο. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τη δομή της έκθεσης. Μπορεί να είχαμε κι άλλες απόψεις δικές μας για τη δομή, αλλά τέτοια ώρα δεν έχει νόημα να πάμε να αλλάξουμε τη δομή. Είναι αυτή που είναι, έχουν υποβληθεί όλες οι τροπολογίες με βάση την ισχύουσα δομή και δεν θα ήταν καθόλου πρακτικό να πάμε να αλλάξουμε τη δομή. Πάει αυτό λοιπόν. Το πιο σημαντικό θέμα για μας είναι να οργανώσουμε τις εργασίες από τώρα και μέχρι την Ολομέλεια με τρόπο τέτοιο ώστε οι ομάδες να μπορούν να συζητήσουν σωστά τις τροπολογίες. Έκανα και κατηδίαν συζήτηση με τον Σαλβαντόρ για αυτό το θέμα και είπαμε ότι θα πρέπει οι προτάσεις 2 Μαΐου για τις συμβιβαστικές τροπολογίες να κατατεθούν, γιατί 3 και 4 Μαΐου θα συνεδριάσει η ομάδα μας και θέλουμε χρόνο μέχρι την τελική ψηφοφορία στην Επιτροπή να συζητήσουμε τις, τροπολογίες αυτές. Και από ό,τι κατάλαβα, ο Σαλβαντόρ μπορεί να δεχτεί την ε, πρότασή μας αυτή και αυτό μας ικανοποιεί ως ομάδα. Συμφωνώ ότι πρέπει να βρεθούν ευρείες λύσεις για κάποια σημαντικά θέματα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στα πάντα, όμως μπορούμε να ε, είμαστε διαπραγματευτές δυναμικοί απέναντι στο Συμβούλιο, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι η πρόκληση μεγάλη είναι στην συνάντηση με το Συμβούλιο κατά την οποία θα ψάξουμε να βρούμε έναν μια αποτελεσματική ε, διαδικασία διαλόγου με τη διαδικασία της σύμφωνης γνώμης. Και αν είμαστε χωρισμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δυσκολευτούμε πολύ περισσότερο να εξεύρουμε καλές λύσεις με το, στο διάλογο με το Συμβούλιο. Οπότε συμφωνώ. Πρέπει να δουλέψουμε τις τροπολογίες και να βρούμε όσο πιο συμβιβαστικές και ευρείες τροπολογίες γίνεται. Βέβαια υπάρχουν όρια. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες αξίες που είναι διαπραγμάτευτες, Αλλά αν να τηρήσω με τα χρονοδιαγράμματα, εγώ συμφωνώ με τις προτάσεις του εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κάρλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν για τη μέθοδο. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Προσβλέπουμε με ενδιαφέρον την κατάθεση των τροπολογιών του εισηγητή, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διαχειριστούμε τις πολλές τροπολογίες και εμείς θα συγκεντρώσουμε τις δικές μας για να τις περιορίσουμε και να τις μειώσουμε κατά 30% διατηρώντας τις αρχικές μας ιδέες. Οι τροπολογίες όμως εξακολουθούν να είναι πάρα πολλές, οπότε θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι. Τώρα για τη δομή της έκθεσης, το μόνο που ίσως ε, θα θέλαμε να αλλάξουμε, να αρχίσουμε με την ε, χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, υπογραμμίζοντας έτσι την ανάγκη να δούμε το ζήτημα των ιδίων πόρων, που υποθέτω ε, ότι υποστηρίζονται ευρέως από το Κοινοβούλιο. Πέρα από αυτό νομίζω ότι είδω μη θα πρέπει να, αποδομεί στην, να αποσκοπεί στην, απο, στην αποστολή ενό μηνύματο προ την Κομισιόν και το Συμβούλιο για τι προτεραιότητέ μα. Ε, την τελευταία φορά που στο Στρασβούργο σα είπα και έχω αυτή την εντύπωση και μελετώντας τις τροπολογίες, δεν θα αναφερθώ και στην κάθε μία, αλλά κοιτάζοντας τις τροπολογίες και τις δικές μας, η πρόκληση δεν ξέρω, δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για προτεραιότητες, γιατί όλα είναι προτεραιότητες έτσι όπως τα έχουμε καταγράψει. Θα είμαι λίγο κοινικός εδώ, αλλά δεν έχουμε αρνητικέ προτεραιότητες. Τα, τα λέω και τα ξαναλέω κάθε φορά βέβαια. Αλλά όλα είναι σημαντικά. Όλα αποτελούν προτεραιότητα τώρα. Δεν λέω ότι αυτό είναι λάθος. Αλλά κάνοντας κάποιους υπολογισμούς θα αυξηθεί μετά από τις προτεραιότητες κατά 30-40% ο προϋπολογισμός. Δεν ξέρω αν είναι αξιόπιστο, οπότε αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, να δούμε δηλαδή ποιες ε, τροπολογίες δίνουν αξιοπιστία στον προϋπολογισμό, γιατί ανάγοντας τα πάντα σε προτεραιότητες ε, δεν θα είμαστε αξιόπιστοι ούτε προς την κοινή γνώμη ούτε προς τα άλλα θεσμικά όργανα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση λοιπόν. Εμείς προσπαθήσαμε να το αναδείξουμε αυτό μέσα από τις τροπολογίες μας, δίνοντας κάποιες κατευθύνσεις, αλλά και άλλες ομάδες είχαν πρωτοβουλίες σε αυτό το τομέα. Εδώ είναι μια κοινή πρόκληση λοιπόν με τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να δείξουμε ότι το αντιλαμβανόμαστε. Όχι ότι λέμε ότι δεν μπορεί να αυξηθεί ο προπολογισμό, αλλά αν χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα, θέλουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες, όχι περιχαρακώνοντας ορισμένα πράγματα από αυτά που κάνουμε με τις αρχικές ε, ε, τροπολογίες, περιχαρακώνοντας δηλαδή κάποια θέματα του προϋπολογισμού, αλλά αναδεικνύοντας προτεραιότητες. Εμείς ε, έχουμε δυνατότητα να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, διαπραγματευόμενοι με τρόπο τέτοιο ώστε στο τέλος να φαίνεται αυτή η προσέγγιση, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε βέβαια να ικανοποιήσουμε όλους τους βουλευτές εδώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να παρέμβω εδώ και να πω ότι η έκθεσή μας θα πρέπει να είναι έκθεση για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε πιο λεπτομερή νομοθεσία και να μπούμε στο βάθος των επιμέρους πολιτικών. Γιατί κάποιες τροπολογίες δίνουν αυτή την εντύπωση. Πάνε να προδικάσουν πράγματα τα οποία έπονται αναγκαστικά. Θα το δούμε αυτό και λεπτομερέστερα, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις κατευθυντήριες γραμμές, όχι λεπτομερή νομοθεσία, αλλά δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτό θα μας βοηθήσει. Ευχαριστώ. Να ξεκαθαρίσω ότι οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες για το συμβιβασμό και όλες οι πολιτικές ομάδες έδειξαν ότι είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν προς τις συμβιβαστικές αυτές λύσεις. Το θέμα του χρόνου όμως εδώ γίνεται κρίσιμο. Έχουμε δύο πράσινες εβδομάδες μπροστά μας και πρέπει παρόλα αυτά να ψηφίσουμε στο τέλος Μαΐου, μετά μια ενδιάμιση εβδομάδα και μετά ψηφίζουμε στην Ολομέλεια. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ομάδες εκτός της Επιτροπής μας να μην νιώσουν ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε από το νου μας και δεν μας ενδιαφέρει η στήριξη της Ολομέλειας. Το θέμα είναι να μας υποστηρίξει η Ολομέλεια με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Είναι λοιπόν κρίσιμο την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει επικοινωνία ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες για τις συμβιβαστικές λύσεις. Γιατί αν οι συμβιβαστικές λύσεις είναι έτοιμες μόνο στις 2 Μαΐου, τότε γνωρίζουμε ότι αυτή την εβδομάδα των πολιτικών ομάδων θα πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις οι πολιτικές ομάδες και κανονικά θα ψηφίσουν στις πολιτικές ομάδες την επόμενη εβδομάδα του Στρασβούργου. Πρέπει να έχει υπάρξει επικοινωνία λοιπόν ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες γιατί αλλιώς ο κίνδυνος της ψηφοφορίες μας στην Επιτροπή μας δεν θα στηριχθεί από την Ολομέλεια που είναι μόνο δύο εβδομάδες μετά. Απαιτείται χρόνος βέβαια για τις συμβιβαστικές ε, προτάσεις. Αυτό το έχουμε πει, το έχουμε παραδεχτεί. Απαιτείται να τις έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας την επόμενη εβδομάδα. Αν καθυστερήσει αυτό για τη Δευτέρα Μαΐου, τότε φοβάμαι ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Αν δεν υπάρξουν ε, ε κάποιες μορφές επικοινωνίας εντατικές ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες την επόμενη εβδομάδα. Τώρα για τη δομή της έκθεσης για μας, όπως και για τους φιλελευθέρους, έχει σημασία να βάλουμε σε ισχυρότερο ε, βάθρο το θέμα των ιδίων πόρων. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία η συζήτηση αυτή. Και αν το Κοινοβούλιο δεν ξεκαθαρίσει τη σημασία που έχουν ήδη οι πόροι στην περίπτωση αυτή, γνωρίζοντας ότι το θέμα έτσι και αλλιώς θα είναι πολύ σοβαρό πολιτικό θέμα συζητήσεις του Συμβουλίου, τότε δεν θα είναι σωστό. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να αλλάξετε τη σύνολη δομή του έκθεσης όπως λένε κάποιοι από το Άλντε, αλλά υποστηρίζουμε ότι κάποιες από τις θέσεις μας για, τις, ε, ή για τους ιδίους πόρους πρέπει να τεθούν στην αρχή της ε, έκθεσης γιατί η, η αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα είναι πολύ σημαντικό θέμα. Τώρα για το μέγεθο του προϋπολογισμού. Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για το περιεχόμενο των μεμονωμένων πολιτικών, αλλά όλες οι πολιτικές ομάδες εξετάζουν σε αυτή τη φάση τις προτεραιότητες και τις λεγόμενες ιστορικά μη προτεραιότητες. Όπως είπα και λίγες εβδομάδες, αν τίποτα δεν αλλάξει στο επίπεδο των NFF, τότε δεν υποστηρίζουμε ούτε αύξηση ούτε μείωση του προϋπολογισμού. Αν εμείς πούμε στην πρώτη παράγραφο της έκθεσης ότι τα βασικά προβλήματα είναι η έλλειψη, η ενέργειας σαν παράδειγμα και άλλα δύο θέματα, φοβάμαι ε, ότι αυτό είναι περιοριστικό για το μέλλον. Θα μπορούσαμε βέβαια να μιλήσουμε για το πρασίνισμα πάρα πολύ εύκολα, γιατί ο καθένας υποστηρίζει ότι πρέπει να πρασινίσουν σε εισαγωγικά πολλές πολιτικές μας, αλλά πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Όταν λέμε ότι πρέπει να πρασινίσουμε την κάψα παράδειγμα, την ΠΑΚ συγγνώμη, ε, τι εννοούμε όταν θέλουμε να κάνουμε τον εξυγχρονισμό της, ε, ε, της κοινή αγροτικής πολιτικής. Τι εννοούμε όταν θέλουμε να εξυγχρονίσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία. Όλα αυτά δεν μπορεί να λείπουν από την έκθεση. Αν λείπουν τότε φοβάμαι ότι εμείς σαν κοινοβούλιο δεν θα μπορέσουμε να πιέσουμε για μια ποιοτική συζήτηση στο Συμβούλιο. Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν ξεκάθαρα τις προτεραιότητές μας και τότε μόνο μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα των ιδίων πόρων και το θέμα της αύξησης του προϋπολογισμού. Μόνο αν πλούσιο, καταστήσουμε πιο πλούσιο το περιεχόμενο της συγκεκριμένης πρότασης. Οι τροπολογίες σχετικές λοιπόν με αυτά τα οποία είπα είναι κρίσιμες για μας και από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα στηρίξουμε την συνολική έκθεση. Έχει σημασία λοιπόν να προχωρήσουν γρήγορα οι συμβιβαστικές τροπολογίες. Το θέλουμε όλες οι πολιτικές ομάδες, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε έγκαιρα την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Διευκρινιστικά. Πολύ σωστά αυτά που λες. Προφανώς όταν συζητάμε το ποσό που θα χρειαστούμε στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, πρέπει να, δούμε, να μιλήσουμε και για την πολιτική που θέλουμε. Για την ΚΑΠ, για παράδειγμα, θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε πράγματα όπως δημόσια κονδύλια για δημόσια αγαθά κλπ. κλπ. Όχι όμως να πούμε ότι οι αγρότες ε, θα πάρουν τόσο τις 100 για αυτό. Στη διαρθρωτική πολιτική πάντα υπήρχαν κάποιες υποδείξεις για τις περιφέρειες και τι έπρεπε να κάνουν ή να πάρουν. Αυτό ενώ όταν μιλάω για νομοθεσία. Γιατί βεβαίως κάποια στιγμή θα τα πιάσουμε και αυτά τα θέματα όλα όταν προχωρήσουμε στους ε, κοινούς κανόνες για την ε, ΚΑΠ, για, τη διαρθρωτική, για την πολιτική συνοχής ε, κλπ. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η δουλειά δεν πρέπει να γίνει εδώ, στην έκθεση ΣΟΥΡ. Η αιρεσιμότητα, οι όροι κλπ, οι γενικές κατευθύνσεις, εντάξει. Αυτά ναι, όχι άλλα. Από το ECR, νομάδα. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ σημαντικά. Γιατί αν στην ομάδα των συντονιστών δεν αποκτήσουμε την υποστήριξη των πολιτικών ομάδων για τις συμβιβαστικές τροπολογίες, τότε πολλές τροπολογίες θα ψηφιστούν στην Ολομέλεια και θα καταλήξουμε να ψηφίζουμε χίλιες ε, τροπολογίες στην Ολομέλεια. Αυτό είναι καταρχήν αντιπαραγωγικό και επίσης θα διατρέξουμε τον κίνδυνο να ψηφίσουμε μια έκθεση χωρίς συνοχή όπου θα ε, περιέχονται πολλά και διάφορα τάκτος ερημένα. Τώρα το δεύτερο, οι ίδιοι πόροι. Ε, δεν ξέρω γιατί πρέπει αυτό να το βάλουμε πρώτο γιατί αν μιλήσω με πρώτα για αυτό το θέμα στην έκθεση. Μπορεί να δημιουργηθεί εντύπωση στην Ευρώπη ότι αυτή δεν είναι μόνο ακαδημαϊκή συζήτηση. Να, να, να μιλήσουμε, να το αναφέρουμε το θέμα και να το ε, εξετάσουμε εμείς ε, είμαστε κατά της ανάπτυξης του θέματος, αλλά το να το βάλουμε πρώτο-πρώτο στην έκθεση θα δώσει την εσφαλμένη εντύπωση ότι αυτό υποτίθεται ότι είναι το μείζον θέμα για τη λήψη απόφασης και αυτό δεν συμβαίνει. Καταλαβαίνουμε τις ε, πολιτικές, ε, τα πολιτικά ενδεχόμενα μια τέτοιας διαδικασίας. δεν θέλω να αλλάξει λοιπόν αυτό. Πώς θα αποφύγουμε όμως συζήτηση για τη μεταρρύθμιση πολιτικών όταν θα μιλάμε για τη χρηματοδότησή τους. Εγώ θέλω να αποφύγουμε να συζητήσουμε τις μεταρρυθμίσεις των πολιτικών όταν μιλάμε για τον προϋπολογισμό, γιατί αυτό είναι δουλειά άλλων επιτροπών. Άλλοι πρέπει να συζητήσουν για τις αλλαγές στην ΚΑΠ και σε άλλες πολιτικές. Έτσι λοιπόν, εάν εισάγουμε, εισαγάγουμε τέτοια ε, θέματα ουσίας στην έκθεση αυτή, είναι επικίνδυνο, είναι ένα ρίσκο. Ένα άλλο ρίσκο είναι να λάβουμε αποφάσεις που εύκολα τεκμηριώνονται ε, στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020, αλλά δύσκολα τεκμηριώνονται βάσει των συνθήκων. Καλύτερα να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου τρόπον την από την πίσω πόρτα θα ε, εισαγάγουμε μεταρρυθμίσεις που δεν εδράζονται στις συνθήκες και που αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις των κρατών μελών μεταξύ τους. Γι' αυτό προτείνω να αναφερθούμε στις σαφείς υποχρεώσεις βάσει των συνθήκων και λιγότερο σε πολιτικά κείμενα ε, από σήμερα το σημαντικότερο είναι να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα ούτω ώστε να σταματήσουμε αυτή τη χιονοστιβάδα της κατάθεσης τροπολογιών στην Ολομέλεια. Ξέρουμε τι γινόταν στο παρελθόν. Η ψηφοφορία θα είναι πολύ δύσκολη, αλλά όσο λιγότερες τροπολογίες χρειαστεί να ψηφιστούν στην Ολομέλεια, τόσο το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Για την ομάδα Ευχαριστώ. Δεν είμαι η εκπρόσωπος στην Επιτροπή ΓΚΟΕ, αλλά δραστηριοποιούμε και ως αναπληρώτρια. Είναι πραγματικά δύσκολο το θέμα. Πρώτα πρέπει να πιάσουμε τα δημοσιονομικά, ταυτόχρονα κάνοντας και συζήτηση για το θέμα της πολιτικής συνοχής και πώς θα συνεχιστεί ως ένα μέρος των δημοσιονομικών. Όλα τρέχουν παράλληλα. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε να έχουμε ισορροπημένη και προσεκτική προσέγγιση και να μην χάσουμε από τα μάτια μας το στόχο περί τίνος πρόκειται. Στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα, όλες αυτές οι πιστώσεις και η χρήση τους πρέπει να συμβάλλουν στην ε, εξισορρόπηση των μεγάλων διαφορών. Ε, εκεί είναι η μεγάλη συμβολή τους. Και αν δούμε και τις γνωμοδοτήσεις άλλων επιτροπών, τι επιθυμίες υπάρχουν. Ε, αν τα δούμε όλα αυτά θα διαπιστώσουμε ότι είναι μεγάλο το δημοσιονομικό μας πρόβλημα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για το συνολικό ύψος και αν αυτό είναι αρκετό για κάποια πράγματα που θέλουμε να κάνουμε ε, στον τομέα της συνοχής για παράδειγμα. Το λέω αυτό διότι υπάρχουν προβληματικές καταστάσεις και προκλήσεις που τα τελευταία 10-20 χρόνια ίσως δεν έπαιξαν τόσο μεγάλο ρόλο όπως παίζουν τώρα γιατί υπήρξαν ανατροπές στον τομέα του περιβάλλοντος. Η φτώχεια επίσης τώρα απέκτησε πολύ μεγαλύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια από ό,τι άλλες προκλήσεις και λόγω της ε, ένταξης νέων μελών. Αυτό εδώ παίζει μεγάλο ρόλο. Αυτά είναι θέματα τα οποία μας προβληματίζουν και εγώ νομίζω ότι είναι λάθος να μιλήσουμε πρωτίστως για τους ιδίους πόρους. Όμως το θέμα των ιδίων πόρων πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγάλη ειλικρίνεια. Είναι θέμα που αντιμετωπίζει πολλές πιέσεις και πολλές φορές ε, τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν προσχηματικά τους ίδιους πόρους για να μην κάνουν κάποια πράγματα. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις ισχυρές και λιγότερο ισχυρές χώρες εδώ. Αυτό που με απασχολεί στο, στην έκθεση Σούρε είναι αυτή η πολύ στενή σύνδεση πολιτικών. Για παράδειγμα, πολιτική συνοχής προς την Στρατηγική Ευρώπη 2020. Νομίζω ότι πολύ προσεκτικά θα πρέπει να ξαναδούμε μήπως αυτό δεν είναι σωστό ή αν είναι. Γιατί έχουμε κάθε τους πολιτικούς τομείς ε, που έχουν ε, προδιαγραφεί στα πλαίσια της ε, στρατηγικής 2020 και αργότερα θα μιλήσουμε για τις οριζόντιες πτυχές της πολιτικής συνοχής. Οπότε αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα συναρθρώσουμε σωστά γιατί δεν είναι επαρκής η παρουσίασή τους με βάση την τωρινή εικόνα και τον πίνακα. Δεν ξέρω, αργότερα μπορεί να χρειαστεί να επανέλθω μετά από τους άλλους συναδέλφους. Και τώρα η Μάρτα Ανδρέασεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αναφέρθηκα ήδη στην δυσκολία που υπάρχει για μακρόχρονο προγραμματισμό όταν περνάμε μια κρίση. Συμφωνώ ότι η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 115 παραγράφους, γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση τόσο λιγότερο αποτελεσματική θα είναι. Σχετικά με το περιεχόμενο της έκθεσης, νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα σχόλια τα οποία έκαναν οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων χτες στην συνάντηση που είχαμε μαζί τους. Δυστυχώς πολλοί από εμά εδώ δεν ήμασταν εκεί. Οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων εξέφασαν την αγωνία τους για την κρίση. Θέλουν να υπάρξει μια αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συγκεντρώσει την προσοχή των προϋπολογισμών στις βασικές προτεραιότητες. Και ιδιαίτερα στο θέμα της απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν εξοικονομήσεις για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση για περισσότερη χρηματοδότηση. Και δεν συζητάμε το θέμα της εξοικονόμησης. Μιλάμε για να βάλουμε τους ίδιους πόρους σαν πρώτο θέμα, αλλά δεν συζητάμε το θέμα της εξοικονόμησης. Ένα άλλο από τα θέματα στα οποία συζητήθηκα χθε είναι το, το θέμα της χρηματοδότησης της συνοχής. Όλοι συμφωνούν ότι δεν υπάρχουν ε, χρήματα για συγχρηματοδοτήσεις και για προγράμματα συγχρηματοδότησης. Οπότε γιατί εμείς ε, ε, μένουμε στο συγκεκριμένο αυτό το τομέα ενώ δεν υπάρχουν πιστώσεις. Τέλος, υπάρχει ο κίνδυνος Ε, δημιουργίας ε, ενός ε, χρηματοπιστωτικού, μάλλον ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα σε πολλούς και θυμούνται την περίοδο του 1980, της δεκαετίας μάλλον του 80. Λοιπόν, διαφωνώ να βάλουμε τους ίδιους πόρους στην πρώτη θέση, διαφωνώ με το να υπάρξει έστω και αναφορά στο θέμα των ιδίων πόρων. Αυτό με, τους, ε, με τη Σουηδία και το αρνητικό παράδειγμα στη δεκαετία του 80 με το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι γνωστό σε όλους. Καμιά φορά όμως ε, ξέρουμε ότι είναι πολύ νωρίς ε, στα πλαίσια μιας διαδικασίας και γι' αυτό παρουσιάζεται αποτυχία ή άλλες φορές γίνεται κάτι υπερβολικά αργά. Γιώραν, σύντομα. Πολύ σύντομα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Θυμηθούμε ότι πρώτα απ' όλα αυτό έγινε σε μία χώρα και αυτή είναι μεγάλη διαφορά αν σκεφτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με το μισό εκατομμύριο Επίσης, ε, πρόκειται για ένα ποσό που ήταν 20 φορές μεγαλύτερο από αυτό το οποίο προτείνεται τώρα, άρα υπάρχει μεγάλη διαφορά των δύο θεμάτων αυτό. Λοιπόν, μιλάει κάποιος πιο ειδικό στο θέμα από ότι είμαστε εμείς. Λοιπόν, αυτό ήταν το γενικό εισαγωγικό κομμάτι, μίλησαν οι εκπρόσωποι των ομάδων, το ΕΛΚ λείπει. Αλλά αν δεν θέλει να πει κανείς κάτι για τα γενικά, μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση στο κομμάτι αυτό. Α, βλέπω μέλη του ΕΛΚ. Γιάνν Γκεμπράντιτ, Τζέιμς Έλλης, Ιβαν και Κωνσταντσε Κρέλ ζητούν το λόγο. Θέλετε να μιλήσετε για το γενικό εισαγωγικό κομμάτι ή για το πρώτο μέρος, δηλαδή τις προκλήσεις και τις προτεραιότητε. Όχι τώρα. Αμέσως, όταν θα μιλήσουμε για τις πολιτικές προτεραιότητες, και τις προκλήσεις. Τότε θα μιλήσουμε για την έκθεση και τις σχετικές με αυτό το θέμα τροπολογίες, τα άρθρα 1 μέχρι 89 στην έκθεση και θα δείτε το πάκο το μεγάλο με τις τροπολογίες είναι 1 με 4. Α, γενικά. Ο Γιάννη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στο τέλος της περασμένης χρονιάς ε, πήγαμε να επηρεάσουμε τις διαπραγματεύσεις και για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Συμβούλιο αρνήθηκε. Για να είμαι ειλικρινής αναρωτιέμαι μήπως στο τέλος καταλήξουμε σε μια έκθεση και που μου φαίνεται προς τα εκεί πάμε ε, που δεν θα ε, είναι σαφής. Ποια θα ήταν η θέση μας στη Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Τώρα συνεχίζονται, μιλάμε για αποφάσεις που θα ληφθούν για το Ταμείο Συνοχής στην γεωργική πολιτική. Αν συμμετείχε κάποιος εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου, τι θα έλεγε. Γιατί δεν έχουμε θέση ως Κοινοβούλιο στα θέματα αυτά. Αν προχωρήσουμε όπως κάνουμε τώρα, έχουμε όλες τις προτεραιότητες στο τραπέζι και αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνουμε θέση τελικά. Είπαμε ότι θα επισέλθουμε στην Επιτροπή αυτή σε επιμέρους ε, πολιτικές, αυτή την Επιτροπή. Κάποιοι λένε όχι, κάποιοι λένε ναι. Ήλπιζα πριν αρχίσουμε να δουλεύουμε σε αυτή την Επιτροπή, ήλπιζα ότι θα έχουμε μια πανοραμική άποψη ως Επιτροπή Δηλαδή μια πανοραμική εικόνα που θα μας επέτρεπε να σταθμίζουμε τη σημασία κάποιων τομέων πολιτικής. Όλοι συμφωνούμε γενικά για τον εξυγχρονισμό, τη σημασία της ε, ε, στρατηγικής 2020, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, η φορεία και όλα αυτά. Αλλά αν όλα αυτά δεν τα μεταφράσουμε σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικών, τότε τι νόημα έχει που έχουμε ένα γενικό όραμα. Ε, δύσκολο είναι να βρούμε το όραμα, αλλά ακόμα πιο δύσκολο είναι να βρούμε την τόλμη να πάρουμε αποφάσεις που θα είναι τα επακόλουθα του γενικού οράματος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα εδώ. Οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες. Αν βρούμε συμβιβαστικές λύσεις που θα βρουν σύμφωνους όλους, στο τέλος θα έχουμε μια θέση που θα είναι μη θέση από πολιτική άποψη και δεν θα μπορέσουμε να ασκήσουμε καμία επιρροή σε όλη τη διαδικασία μέχρι το τέλος της, μέχρι να συμφωνήσει το Συμβούλιο για το Μελλοντικό Πολιετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το MFF. Θα πρέπει να υπογράψουμε απλώς μια τελική συμφωνία και τίποτα παραπάνω. Πρέπει λοιπόν τις επόμενες εβδομάδες να κοιτάξουμε να πιεστούμε, να βρούμε όχι μόνο ε, τροπολογίες που θα βρίσκουν σύμφωνους όλους, αλλά να κάνουμε επιλογές. Οι επιλογέ σημαίνει ότι δεν θα συμφωνήσουν όλοι. Καλύτερα όμως να έχουμε ισχνή πλειοψηφία, η οποία όμως θα επιτρέπει να κάνουμε πολιτικές επιλογές και έτσι θα έχουμε μια στεναρή πολιτική θέση απέναντι στο Συμβούλιο, παρά να έχουμε μια θέση όπου θα συμφωνούν όλοι, αλλά δεν θα κάνουμε πολιτικές επιλογές. Αυτό πρέπει να δούμε τις επόμενες εβδομάδες και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες που δεν θα είναι αποδεκτές από όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξη. Νομίζω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε μια έκθεση η οποία θα λέει κάποια πράγματα. Και επίσης θα έχουμε μια αρκετά ικανοποιητική πλειοψηφία πίσω από την έκθεση και θα βεβαίως θα πάρουμε αποφάσεις, δεν θα τα βγάλουμε πέρα μόνο μέσα από συμβιβαστικές τροπολογίες, πρέπει και να αντιπαρατεθούμε. Αλλά αν ως κοινοβούλιο δεν πάρουμε θέση, τότε θα μας κάνει το Συμβούλιο ό,τι θέλει. Και γι' αυτό και για λόγους ε, ε, ε, επιβίωσης και αυτοσυντήρησης πρέπει να πάρουμε θέση. Η γενικά. Ο Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Στην τελευταία συνάντηση συνδιάλεξη με το Συμβούλιο δεν καταλήξαμε πουθενά για τις ιδίους πόρους. Δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε συμφωνία. Η πρότασή μου, λοιπόν, χωρίζεται σε δύο μέρη. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την ε, να αντιδράσουμε σε αυτή την πρόταση που κάνει το κράτη-μέλη. Να παγώσουμε στο επίπεδο του 2013 το κοινοτικό προπολογισμό. Ε, συμφωνήσαμε να πούμε όχι, διότι σε αυτή την περίπτωση, εάν συμφωνήσετε είναι θέμα. Αν δεν το συμφωνήσετε και θέλετε ένα νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, πρέπει να δικαιολογήσουμε πώς βρίσκουμε τους πόρους. Τώρα, υπάρχει και η άλλη δυνατότητα της χρηματοδότησης των ιδίων πόλων, όχι με αύξηση ε, των φόρων, με αύξηση του ΦΠΑ και ένα άλλο παράδειγμα από χθε που μας απέδειξε ότι δεν είναι εντελώς λαθασμένο το σύστημα. Τα κράτη-μέλη στο Κανκούν συμφώνησαν για κάθε χρόνο να διαθέτουν 2,4 δις για να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές αλλαγές. Χθες στην Επιτροπή Προπολογισμών είχαμε μεγάλο πρόβλημα, διότι είπε ο εισηγητής γιατί θα πρέπει να πληρώνουμε εμείς για να κάνουν κόλπα οι Κινέζοι και οι άλλοι. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε μία απάντηση σαφή. Ή διαφωνούμε κάθετα ή συμφωνούμε με τις χώρες που έχουν την πλειοψηφία συμβούλιο. Τις σκανδιναβικές χώρες, την Γερμανία που έκαναν αυτή την πρόταση, που έβαλαν αυτή την πρόταση γραπτός. Ευχαριστώ. Κωνσταντζε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ ήθελα να πω δύο λόγια για τη γενική συζήτηση. Συμφωνώ ότι στην έκθεση του κυρίου Καρίγκα πρέπει να δώσουμε γενικές κατευθύνσεις για αλλαγές στους τομείς των πολιτικών, αλλά δεν μπορούμε να αρχίσουμε να νομοθετούμε. Άλλωστε, δουλειά μας είναι και αυτή και θα καταπιαστούμε αργότερα με τις λεπτομέρειες ξέρω ότι όταν επισέλθαμε σε επιμέρους νομοθετήματα πάμε σε μεγαλύτερο βάθος και αυτό το βλέπω από άλλες επιτροπές. Θα γίνει πολιτική αντιπαράθεση στις καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές και η απόφαση θα γίνει στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης. Δεν μπορεί δηλαδή εδώ να πάμε ε, μέσα από μια ταχεία διαδικασία δεν μπορεί δηλαδή να πιστεύουμε ότι μέσα από την έκθεση αυτή στα γρήγορα, στην ΚΑΠ, στην πολιτική συνοχή θα βρούμε γρήγορες λύσεις για τον εξυγχρονισμό. Πρέπει να τα πιάσουμε με τη σειρά. Ο κ. Γκαρίγα έκανε καλές προτάσεις, ιδιαίτερα στην πολιτική συνοχή. Δηλαδή, πάμε αρκετά σε βάθος για να δώσουμε κάποιες προδιαγραφές για αργότερα, για το πώς θα διαμορφωθεί η νομοθεσία καλά. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την γενική συζήτηση. Θες να κλείσεις το κομμάτι αυτό, Σαλβαντόρ. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Εάν όντως οι πολιτικές ομάδες θέλουν να έχουν στα χέρια τους ο συντομότερο εδώ τις συμβαστικές τροπολογίες, ίσως θα πρέπει ο εισηγητής να επιταχύνει τη δουλειά που θα κάνει με τη συνεργασία της ε, γραμματείας. Είπαμε ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τις ημερομηνίε τι οποίε θα μπορούσα εγώ να συναντηθώ με τη γραμματεία πολύ νωρίτερα από ό,τι είχε προβληθεί. καταρχά για να μπορέσω να έχω έτοιμε τι συμβαστικέ τροπολογίε και να τις αποστείλω το συντομότερο δυνατό στις πολιτικές ομάδες. Όσον αφορά την ουσία του όλου θέματος, μένω παρά το γεγονός ότι τώρα θα μπούμε για τα πιο σημαντικά θέματα στις απόψεις των πολιτικών ομάδων. Αλλά καταρχήν θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι η ιδέα που μας οδήγησε και η δομή αυτής της έκθεσης είναι να κάνουμε μία πολιτική διακήρυξη. Και απευθύναμε σε δύο λαμπρούς νέους συναδέλφους, τον Θέλ Μπράντι και τον Μπάς. Τελικά πρέπει να πω το εξή. Θα πρέπει να είμαστε, να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε. Μέσα της Επιτροπής μας, τη ΣΟΥΡ, μπορούμε να προσπαθήσουμε να μεταβάλουμε τις κοινοτικέ πολιτικές. Αλλά πιο έμπειροι κοινοβουλευτικοί συνάδελφοι από μένα, η κυρία Κλέρ που μόλις τώρα πήρε το λόγο μας είπε ότι οι αρμόδιες επιτροπές θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν. Εγώ μπορώ να υποβάλω μια πρόταση η οποία πραγματικά να είναι επαναστατική και ριζοσπαστική σε σχέση με τις προτεραιότητες και να αποτελεί πραγματική τομή σε σχέση με τις προτάσεις για τον προπολογισμό, αλλά είμαι σίγουρη ότι στις αρμόδιες επιτροπές δεν θα επιτευχθεί για μια τέτοιου είδους έκθεση καμία συμφωνία. Αυτό το ξέρουμε εκ των προτέρων. Άρα η δική μου η προσέγγιση να φαίνεται κάπως απογοητευτική όσον αφορά του βραχυπρόθεσμους αντικειμενικού στόχου. αλλά πιστέψτε με ότι αν θέλουμε να δώσουμε ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι η μόνη εναλλακτική λύση είναι να λάβουμε υπόψη και τα μελήματα και τις απόψεις των Ορμοδίων επιτροπών. Εγώ δεν βλέπω πώς θα μπορούσα να ενεργήσω διαφορετικά. Και στα πλαίσια αυτών των περιορισμών, οι πολιτικές ομάδες, η Γραμματεία και εγώ προσπάθησαν να, να συντάξουμε μια έκθεση που μπορώ να θεωρήσω την αρκετά καινοτόμο. Όταν θα πρέπει να ψηφίσουμε, ήθελα να έχουμε κατά νου την έκθεση του Συμβουλίου για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Και θα δούμε εάν ε, είναι πολύ ε, διαφορετικές από τις δικές μας, πώς θα ψηφίσετε, αν τις καταψηφίσετε τις προτάσεις αυτές του Συμβουλίου. Και θα δω αν μπορούμε εμείς ε, να καταψηφίσουμε τις προτάσεις του Συμβουλίου θα μπορούσαμε, επαναλαμβάνω, να κάνουμε μια πολύ ριζοσπαστική πρόταση. Το θέμα είναι πώς θα ψηφίσουμε την ώρα της αλήθειας και μπροστά στο Συμβούλιο να μπορέσουμε να λάβουμε τις πραγματικές πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή, αν η τελική πρόταση του Συμβουλίου είναι συμβατή με τη δική μας πρόταση, με την πρόταση Επιτροπής ΣΟΥΡΕ, έχει καλώς. Θα υπερψηφίσω την πρόταση για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικέ. Ιδάλλως θα την απορρίψουμε. Έχουμε τέτοιου είδου εμπειρίε στο παρελθόν. Αλλά θα πρέπει να δούμε και να δώσουμε το, πώς θα δώσουμε το κατάλληλο μήνυμα και μέχρι πού μπορούμε να πάμε σε σχέση με το Συμβούλιο. Αυτά μπορώ να πω προς το παρόν, κυρία Πρόεδρε. One question, bitte. Ερώτηση για τον κύριο Γαρίγκα. Πολύ εκτιμώ την πείρα του και πώς κινείται με τη δική σας προσέγγιση. Γιατί δεν πήραμε όλες τις γνωμοδοτήσεις των ειδικών επιτροπών να τις κάνουμε ένα συμπίλημα και να κάνουμε έκθεση. Τι ρόλο παίζει η Επιτροπή Σούρε. Κάποιο ρόλο παίζουμε κι εμείς. Ο ρόλος μας είναι να δούμε τις γνωμοδοτήσεις των ειδικών επιτροπών και να βγάλουμε ένα γενικότερο συμπέρασμα. Ερωτώ λοιπόν, να κάνουμε ένα συμπίλημα των γνωμοδοτήσεων που υπάρχουν και να τελειώσουμε και να τελειώνουμε. Ναι, δηλαδή όπως στο, στο γάμο, όπου το ζευγάρι συζητάει για τις σχέσεις τους. Αυτά τα είπαμε στην αρχή. Ο, ο Πρόκειται για την προσθέμενη αξία της ΣΟΥΡΕ. Αυτό είναι το μέσο που θα χρησιμοποιήσω για να αναλύσω τις προτάσεις των αρμοδίων επιτροπών. Βεβαίως, εάν δείτε την συνεισφορά κάθε επιτροπής και δείτε την το τελικό σχέδιο εκδόσης θα δείτε ότι δεν παραθέσαμε όλες τις γνωμοδοτήσεις, πήραμε κάποια κομμάτια αλλά προσπαθήσαμε να τις τροποποιήσουμε και να τις προσαρμόσουμε στην γενική δομή σύμφωνα με τις ιδέες και του εισηγητή και των πολιτικών ομάδων. Άρα αυτή δεν είναι η καλύτερη λύση, δηλαδή να προσαρτήσουμε όλες τις ε, ε γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό κορμό στον οποίο θα ενσωματώσουμε τις συνεισφορές, αλλά όχι όλες. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να μπορέσουμε να σωματώσουμε κάποιες ιδέες, αλλά δεν ε, προσθέσαμε τις διάφορες συνεισφορές. Γιατί αν το κάναμε θα ήταν εντελώς διαφορετικό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Τώρα λοιπόν έχουμε θέσει το γενικότερο πλαίσιο και προχωρούμε στη συζήτηση των τροπολογιών μας. Σας είπα ότι η παράγραφη 1 με 89 της έκθεσης είναι η βάση τώρα για τη συζήτησή μας και τα πρώτα τέσσερα πακέτα τροπολογιών. Έχω τρεις ομιλητές στον κατάλογό μου μέχρι τώρα. Δεν κάνουμε γύρω των ομάδων. Όποιος θέλει θα πρέπει να ζητήσει το λόγο. Ο Κάρδι είναι στον κατάλογο ήδη, η Μαρία Καβάλιο, Ιβάιλο Κάλφιν και Καρλ Χακλούντ. Αρχίζουμε, Μαρία. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. The group of amendments that have been discussed and supported by the members of the Έχω καταθέσει τις τροπολογίες που υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Καλύπτουμε κάποιους τομείς σχετικά με την πιθανότητα αύξησης των πιστώσεων για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο στον τομέα της καινοτομίας. Για να προωθήσουμε επίσης και τις βέλτιστες δυνατές επιδόσεις των επιχειρήσεων Uh, of the framework program, of the existing framework program, the seven framework program. So some of the new member states... Νομίζω ότι κάποια από τα κράτη-μέλη σε σχέση με την σημερινή συγκυρία αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα και η κατανομή των πιστώσεων δεν είναι η, η βέλτιστη δυνατή. Παρ' όλα αυτά, επιδόσεις ε, εξαιρετικού επίπεδου υπάρχουν από πάρα πολλές ε, ε, επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες. Um, this was approved yesterday Η πορεία λοιπόν προς την αριστεία η πορεία προς την αριστεία νομίζω θα πρέπει να τονωθεί ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό έχουμε βάλει τις τροπολογίες αυτές που έγιναν δεκτές στην Επιτροπή Ήτρε με μεγάλη πλειοψηφία. Για τη βιομηχανία έχουμε καταθέσει επίσης τροπολογίες για τη στήριξη καινοτόμων και ανταγωνιστικών ε, επιχειρήσεων. Έχει τεθεί επίσης το θέμα της απλοποίησης ε, της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως επίσης και το θέμα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού τομέα. Στον τομέα της ενέργειας είπαμε ότι υπάρχει θέμα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της χρήσης της ενέργειας και να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε πρόσβαση σε καθερή ενέργεια για όλους. Τίθεται το θέμα της χρηματοδότησης και άλλων προγραμμάτων όπως τα διαφθρωτικά Πρέπει πάντως να γίνουν δεκτές ελπίζω οι τροπολογίες που αφορούν την ανταγωνιστικότητα. Για τα οριζόντια θέματα ζητάμε να υπάρξει μια απλούστευση των διοικητικών κανόνων για τα θέματα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα η Ευρώπη θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ, και πιο απλή. Ευχαριστώ, Ιφάιλο. Uh, uh, Ευχαριστώ, Ιούτα. Να κάνω κάποια σχόλια γενικά. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες όμως, γιατί ως ομάδα έχουμε υποβάλει έναν αριθμό τροπολογιών και μονομένα μέλη της ομάδας κατέθεσαν τροπολογίες. Και όταν αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στο κείμενο, θα δούμε τα κείμενα αυτά ε, συγκεκριμένα. Γενικά τώρα για τις αλλαγές των πολιτικών μας, τις πολιτικές προτεραιότητες ε, και το ρόλο του προϋπολογισμού, που είναι αυτό το κομμάτι του έκθεση του Σαλβαντόρ. Όταν μιλάμε για προϋπολογισμό πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ε, τον αντίκτυπο. Σε αυτό το στάδιο όχι να μιλάμε για χρήματα. Βέβαια έχουμε τους περιορισμούς του προϋπολογισμού. Αν αρχίσουμε από τους περιορισμούς, αντίστροφα δηλαδή, φοβάμαι πολύ ότι δεν θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε σωστά τις πολιτικές και τους στόχους που πρέπει να έχει αυτό το δημοσιονομικό μέσο. Πρέπει επίσης να συνδυάσουμε τη σταθερότητα των υφισταμένων πολιτικών και στόχων με την εισαγωγή των νέων προκλήσεων που βλέπουμε ότι θα αναπτυχθούν ε, στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εδώ να αλλάξουμε όλες τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον, είναι ανέφικτο. Δεύτερον, πρέπει να ε, να θυμόμαστε ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα μέσο για να επιτύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε εθνικούς προϋπολογισμούς, έχουμε πρόσθετα συμπληρωματικά δημοσιονομικά μέσα και μηχανισμούς, έχουμε άλλες δυνατότητες, συμπράξη ιδιωτικού δημοσίου τομέα κλπ. κλπ. Δεν θα βρούμε μια-δυο προτεραιότητες και θα πούμε αυτά θα ε, καλύπτονται και θα εξαρτώνται από τον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Πάμε λοιπόν να ε, κάνουμε μια βελτιστοποίηση, να αντιμετωπίσουμε τις προτεραιότητες και να κινηθούμε σε οριζόντιο επίπεδο. Πρώτον, πρέπει να δημιουργήσουμε όλε τι προποθέσει και του όρου για να εφαρμόζεται η συνθήκη τη Λισαβόνα. Γιατί εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα με τη σωστή εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Δεύτερον, η στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Δεν την ξανακάνουμε την πολιτική, υπάρχει. Θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο προϋπολογισμός σε όλους τους τομείς για να δώσουμε τα αποτελέσματα που θέτει η στρατηγική 2020. Να σκεφτούμε τις προτεραιότητες του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου και σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Λέγαμε ότι πολλές χώρες ε, θα εξακολουθούν να έχουν λιτότητα στον προϋπολογισμό τους. Παράλληλα όμως αναμένουμε μεγέθυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας το ίδιο χρονικό διάστημα. Για τη μεγέθυνση χρειάζονται πρόσθετες επενδύσεις. Δεύτερον, έχουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο, έχουμε την οικονομική διακυβέρνηση κλπ. κλπ. Πώς θα ενταχθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στον καλύτερο αυτό οικονομικό συντονισμό. Και αυτό είναι κάτι που θέτει ένα πλαίσιο. Τρίτο, Μιλάμε για μεγαλύτερη σύγκληση των εθνικών οικονομιών. Πώς μπορεί να παίξει ρόλο ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για εδώ. Επίσης, Μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, έρευνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις. Αυτό είναι το πλαίσιο. Εκεί θα βάλουμε τις πολιτικές μας. Σε όλα τα κεφάλαια. Πρέπει να κάνουμε τις ε, απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να κάνουμε δαπάνες στον προϋπολογισμό που θα προσανατολίζονται περισσότερο προς τα αποτελέσματα. Θα πρέπει, ε, μιλάμε για δημόσιες δημόσια κονδύλια για δημόσια αγαθά που δημιουργούν ε, ε, ενεργητικό στην κοινωνία. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν μπορεί επίσης να αγνοεί τις κοινωνικές πτυχές της ευρωπαϊκής εξέλιξης. Απασχόληση, δημιουργία θέσεων εργασίας, αντιμετώπιση των ευάλωτων, το ΜΜΕ, ε, κοινωνικός αποκλεισμός. Βέβαια δεν μπορεί να λύσει όλα αυτά τα θέματα ο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αυτά είναι πρωταρχικά εθνικά θέματα, αλλά δεν μπορούμε και να τα αγνοεί ο ευρωπαϊκός προπολογισμό. Έχουμε σαφείς προτεραιότητε και φαίνονται και χαίρομαι γι' αυτό στις διάφορες προτάσεις. Έρευνα και ανάπτυξη που πρέπει να είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μα. Ενέργεια, εξωτερικέ πολιτικέ κλιματική αλλαγή, βιοπικιλότητα, υποδομές μεταφορών, ε, διάστημα, νεολαία, νεότητα, ε, θαλάσσια πολιτική κλπ. Επίσης, ε, για λίγα λόγια για κάποια θέματα που πρέπει επίση να συζητηθούν. Όταν μιλάμε για τον προπολογισμό, θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι δυνατότητε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα χρηματοδοτικά μέσα και να δημιουργήσουμε μόχλευση για τον προπολογισμό δεν έχω καταλάβει ε, τι εννοούν οι συνάδελφοι που μιλάνε για αρνητικές προτεραιότητες. Να το πούμε καθαρά. θέλουμε περικοπές. Ποιο θα λάβει την απόφαση, γιατί υπάρχουν διάφορες αποφάσεις που θα ληφθούν από το Συμβούλιο, από το Κοινοβούλιο κλπ. Τέτοια ορολογία, όπως οι αρνητικές προτεραιότητες, δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση στον προπολογισμό κατά τη γνώμη μου. Τρίτον, ευελιξία ό,τι και να αποφασίσουμε για τον προπολογισμό πρέπει αυτό να είναι ευέλικτε, ούτω ώστε να αντιμετωπίζουμε τι νέε προκλήσει που αναπόφευκτα θα ανακύψουν την περίοδο αυτή. Τέλο, υπάρχει ένα θέμα που το έχουμε καταπιαστεί στι τροπολογίε μα. Έχουμε τεράστιο ε, χάσμα μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών που αυξιάνει και θα πρέπει να το δούμε. Έχει να κάνει με τα ρέστα τα ράλς, δεν θα αυξήσουμε τα κονδύλια του προπολογισμού, αλλά με τα χρηματοδοτικά μας μέσα, τα δημοσιονομικά, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει και να έχουμε καλύτερη σχέση μεταξύ υποχρεώσεων και πληρώμων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα καλωσορίσουμε και το συντονιστή από το οποίο ήρθε από τις άλλες του δουλειές. Καλώς ήρθατε. Ενημερώνετε τώρα για το τι συζητήσαμε μέχρι τώρα. Όποτε θέλει, αν θέλει, ναι, να το γράψω το όνομα για να παρέμβει. Κάρλ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σχολιάσω κάτι για τις ε, αρνητικές προτεραιότητες. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα και το θέμα είναι σε ποιο επίπεδο λεπτοπεριών μπορούμε να μιλήσουμε για τις αρνητικές προτεραιότητες. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να πούμε ότι υπάρχει σημεία. Ότι με ευφύ τρόπο θα πρέπει να ελέγχουμε τις ε, δαπάνες για να μπορέσουμε να προσθέσουμε ε, να, κάνουμε μία, ε, να δώσουμε προσθέμενη αξία, να δούμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε οικονομίες, διότι αν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να το κάνουμε με αξιόπιστο τρόπο. Και πρέπει να πούμε ότι εκτός από τις οικονομίες χρειαζόμαστε και περισσότερο χρήματα, περισσότερα κονδύλια. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε, για να το κατορθώσουμε αυτό, ποιε είναι οι παρούσε δαπάνε, για να δούμε πώ μπορούμε να παρέμβουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι βασική αρχή όταν θέλει κανεί να δει πώ θα δημιουργήσει ε, νέα κονδύλια στην, σε ένα προβλήμα στη χρηματοδότηση. Αυτή λοιπόν θα πρέπει να είναι και μία από τις προσεγγίσεις της έκθεσης. Όσον αφορά κάποιες τροπολογίες, σύντομα θα ήθελα να μπορέσω εγώ να σχολιάσω κάποιες από τις δικέ μα τροπολογίες. Από ό,τι κατάλαβα θέλετε πρώτα να συζητήσουμε τις πρώτε 89 παραγράφου. Όσον αφορά το επίπεδο των δαπανών. Τροπολογήσαμε την παράγραφο που αναφέρεται στο 1% των δαπανών. Είπαμε ότι βλέπουμε με όλες τις υποχρεώσεις από τις νίκες Λισαβόνης και τις ε, προτεραιότητες θα πρέπει σήμερα να μπορέσουμε, να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα με το επίπεδο των δαπανών που έχουμε. Και αν θέλουμε περισσότερα χρήματα θα πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι. Θα πρέπει να δούμε αν λοιπόν κάτι τέτοιο είναι δυνατόν ή όχι. Αν δεν είναι δυνατόν δεν είναι. Συγχρόνω. Προσπαθήσαμε να δούμε σε ποιο επίπεδο δαπανούμε. Και εδώ μιλάμε το τι ακριβώς γίνεται με την ε, ε, υπηρεσία εξωτερικών, εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε πώς θα πρέπει γίνουν και οικονομίες στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορέσουμε γενικότερα όλοι μαζί να ενεργήσουμε για να εξοικονομήσουμε χρήματα και να μην ακολουθήσουμε 27 διαφορετικά συστήματα. Προσπαθήσαμε λοιπόν αυτό να το υπογραμμίσουμε και είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε στο Συμβούλιο. Διότι εύκολα φτάνουμε σε μια κατάσταση ώστε την οποία δημιουργούμε μια υπηρεσία για να εξοικονομήσουν ε, χρήματα τα κράτη-μέλη, μετά δεν γίνεται κάτι τέτοιο και δαπανούμε τα διπλά. Τώρα, Είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερους πόρου για την έρευνα και την ανάπτυξη. Είναι πρωταρχικής σημασίας για την ΚΑΠ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μπορούμε να συζητήσουμε εάν θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες περικοπές και περιορισμένες. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα κονδύλια που δαπανώνται για την ΚΑΠ ε, έχουν προθεμένη αξία. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε εκεί τι γίνεται και ε, να δούμε σωστά ποιε είναι οι περικοπές της ΚΑΠ. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε και στην ΚΑΠ ε, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Επίσης, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάπτυξη θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται και πώς θα μπορέσουν κάποιες δαπάνες να τι αναλάβουν τα κράτη-μέλη. Σε θέματα διοικητικά κάνουμε κάποιες προτάσεις εξοικονόμησης. Ξέρω ότι όλοι δεν είναι υπέρ, αλλά είναι σημαντικό δείξουμε ότι αν εξετάζουμε τις διάφορες διοικητικές δομές και είμαστε προσεκτικοί, νομίζω ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα. Δεν είναι συμβολικές ε, οι οικονομίες που θέλουμε να κάνουμε. Και αναφέρομαι, Φερρυπίν, στις ε, τρεις έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εδώ έχουμε συμπληρωματικές δαπάνες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικές οικονομίες. Και αυτό είναι κάτι που αφορά την ε, όλη συζήτηση γιατί είναι διοικητική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι είναι ευαίσθητο το θέμα, αλλά αν θέλουμε να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ξέρω ότι για πολλούς τα πράγματα είναι ε, δύσκολα. Τώρα για τα διάφορα κεφάλαια. Νομίζω ότι θα θέλαμε να έχουμε ένα για την Ευρώπη το 2020, ένα για την διοίκηση και ένα για την εξωτερική πολιτική. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τον θέμα των δαπανών με ευελιξία, διότι ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση και προσβλέπουμε ε, συζήτηση για να μπορέσουμε να τα διαπραγματούμε αυτά και με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ. Ωραία. Οι ιδέες της ομάδας των φιλελευθέρων σχετικά με τη... Ναι, μια έδρα του Κοινοβουλίου, ένας χώρος σε ένα σημείο για όλους τους οργανισμούς, ένα σημάζεμα. Αυτό είναι καλό, γιατί προτρέπουμε και το Συμβούλιο να δει τι μπορεί να κάνει. Βέβαια δεν ξέρω αν θα έχουμε απόλυτη πλειοψηφία, αλλά ακόμα και αν το είχα, την είχαμε στο Κοινοβούλιο, δεν βλέπω πώς θα πιστεί το Συμβούλιο. Όμως, εμείς μπορούμε να του πούμε ότι αυτές οι δαπάνες είναι δικές σας, δεν είναι δικές μας. Ευχαριστώ πολύ, Γιούτα. Κύριος Κλούτε. Και εμείς καταθέσαμε κάποιες τροπολογίες, κάποιες ως γκουε, άλλες από μεμονωμένα μέλη μας. Δεν θα υπησέλθω σε όλα αυτά. Μόνο δύο-τρία θέματα θα θίξω που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά. Μεταξύ άλλων το πρόβλημα της δημογραφικής εξέλιξης που αναφέρεται σε ορισμένα σημεία. Είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν είναι μόνο θέμα κόστους αυτό. Πρέπει να το δούμε. Υπάρχουν κάποιες ε, αλλαγές ε, αναμφισβήτητα, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι οι συντάξει αποτελούν, συνιστούν και αγοραστική δύναμη, που δεν είναι αμεληταία και η γύρανση του πληθυσμού αποτελεί και ένα δυναμικό για ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας. Έχουμε σχετική τροπολογία, μην το ξεχνάμε αυτό. Ε, βέβαια από την άλλη είναι το θέμα της ε, ε, κατανομής και... αλλά μην ξεχνάμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν εδώ για δημιουργία καλών θέσεων εργασίας. Είναι και κομμάτι της στρατηγικής 2020, την ανάπτυξη καλών θέσεων εργασίας βιώσιμων. πολέμηση της φτώχειας και αυτό είναι μια θεματική στη στρατηγική 2020 Πέρσι ήταν και ε, το έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, οπότε αναδείχθηκε σε προτεραιότητα και πρέπει εδώ τώρα να αποκτήσει σάρκα και οστά με συγκεκριμένα μέτρα, να μην είναι ε, ρητορικό το ζήτημα, να αποκτήσει υπόσταση και να καταλάβουν, να ε, νιώσουν οι πολίτες της Ένωσης τι μπορεί να τους προσφέρει και σε αυτό το τομέα, όχι μόνο δηλαδή βιομηχανία και έρευνα, πρέπει και οι πολίτες να πάρουν συγκεκριμένα μηνύματα και να το αισθανθούν αυτό το πράγμα ότι και για μας είναι ε, προστιθέμενη αξία η Ένωση. Ενέργεια, σημαντικό για μας, ε, είδαμε μετά τη Φουκουσίμα που βρίσκονται τα προβλήματα. Στην ενεργειακή πολιτική οπωσδήποτε υπάρχει ε, προτεραιότητα, δηλαδή αλλαγή στους τομείς ενέργειας αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μπορούμε να το δούμε σε επίπεδο εθνικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει εδώ μεγάλη ευθύνη αλλά και μεγάλη ευκαιρία να δει εδώ και να εντοπίσει την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα τελευταίο θέμα που μας ενδιαφέρει πολύ είναι η σταδιακή κατάργηση, το phasing out. Υπάρχουν κάποιες περιφέρειες που εξαιρούνται σταδιακά από το Ταμείο Συνοχής μεταξύ άλλων περιοχές στην Ανατολική Γερμανία που σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από πληρωμές από το Ταμείο Συνοχής. Οι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι αλλάζουν τα πράγματα, ότι υπάρχει μια μετατόπιση προς την κατεύθυνση των νέων κρατών μελών, αλλά υπογραμμίζω και πάλι ότι για να περάσει σε πολιτικό επίπεδο η απόφαση αυτή θα πρέπει να κινηθούμε σταδιακά και να μην έχουμε φνίδιες αλλαγές. Έχω την εντύπωση όμως ότι συμφωνούν και, άλλα κόμματα, και τα άλλα κόμματα εδώ. Υπογραμμίζω απλώς ότι είναι σημαντικό το θέμα και ότι αυτές οι αλλαγές στην πολιτική μας θα πρέπει να μπορούν να απορροφώνται από την κοινωνία. Αυτά. Έχουμε θίξει και κάποια άλλα θέματα, αλλά θα επανέλθουμε όταν μιλήσουμε για τις επιμέρους τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, για την περιφερειακή πολιτική ισχύει αυτό ότι δεν ξέρω κόμματα και πολιτικές ομάδες, ξέρω μόνο τις περιφέρειες. Το λέω λίγο ηρωνικά αυτό, αλλά πραγματικά στο σημείο αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι και νυφάλιοι στην προσέγγιση μας. Ράι Μάρα. Εδώ μιλάμε για τις ε, κύριες ε, προκλήσεις, τις προτεραιότητες, αλλά όχι ακόμα για τη δομή του προϋπολογισμού, το λέω διευκρινιστικά, γιατί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών μιλήσαμε για ε, το προϋπολογισμό και τις διαπραγματεύσεις που μπορούμε να ολοκληρώσουμε ή όχι μέχρι τον Ιούλιο. οι σκιώδεις που μίλησαν στην Επιτροπή Προπολογισμών ζήτησαν εντατικές συνομιλίες για την ευελιξία. και ε, δεν τα καταφέρουμε, υπάρχει μια προθεσμία για να συμφωνήσουμε ή όχι. Αν ε, μέχρι το καλοκαίρι γίνουν δεκτά κάποια αιτήματα, θα πρέπει να δούμε τι ε, επηρεάζεται αρνητικά στον προϋπολογισμό και μετά σε επόμενο βήμα θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Και έτσι ίσως ε, καταλάβει και το Συμβούλιο ότι το συμφέρει να κινηθεί προς κάποια θετική κατεύθυνση. Βέβαια έτσι θα είναι και οι εργασίες μας δημιουργικές. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περιμένουμε Ε, πολλά να κινηθούν, μεταφορά μη σών ε, πιστώσεων ε, και είναι σημαντικό να συμφωνήσει και το Κοινοβούλιο εδώ. Ήθελα απλώς να τα συνοψίσω όλα αυτά για να ξέρουμε και εμείς ότι είμαστε ενωμένοι σε μια γραμμή πλεύσης. Συμπληρώνω ότι και εμείς καταθέσαμε πολλές τροπολογίες και ως ομάδα και με μονομένα μέλη μας ε, αναφέραμε ε, αρκετά θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, τις αρνητικές προτεραιότητες. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες γιατί κάναμε και μια μεγάλη συζήτηση ε, στην ομάδα. Τώρα για τις τροπολογίες μου πιστεύω ότι είναι σημαντικό εκτός από τη στρατηγική 2020 να καταστήσω με σαφές ότι η συνθήκη καθ' αυτή είναι το βασικό σημείο αναφοράς για τις προτεραιότητες στα πλαίσια της δημοσιονομικής πολιτικής, γιατί ε, από τη συνθήκη ε, έχουμε αναλάβει κάποιες πολιτικές υποχρεώσεις, κάποια καθήκοντα και πολλές φορές το Συμβούλιο ε, δεν είναι συνεπές σε όλα αυτά όταν συζητάει για ποσά στα πλαίσια ενός πολιετούς δημοσιονομικού σχεδιασμού. Είναι σημαντικό λοιπόν το θέμα και επίσης όλη η συζήτηση για τη σημασία των επενδύσεων των δαπανών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί θα πρέπει να έχουμε εξοικονομήσεις ή συνεργιστικά αποτελέσματα, συνέργειες και σε εθνικό επίπεδο. Και αυτά πρέπει να τα δούμε πιο εντατικά στο μέλλον, γιατί ε, στο παρελθόν σημειώθηκαν κάποια ελλείμματα στην ανάληψη δράσης. Επίσης ε, πρέπει να δούμε τις ε, γενικές συνολικές πολιτικές προτεραιότητες στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 και των εθνικών προϋπολογισμών, επίσης ε, καινοτόμοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, το συζητήσαμε και αυτό, και τον ευρωπαϊκό, τον ενωσιακό προϋπολογισμό που πρέπει σε τελευταία ανάλυση να χρηματοδοτεί τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Και θα πρέπει να δούμε τι χρειάστηκε στο παρελθόν να, χρηματοδοτηθεί εκτός προϋπολογισμού. Η Γραμματεία έχει καταρτήσει και ε, στοιχεία για τις διμερείς συνεργασίες στον τομέα της έρευνας 5 δις ε, εκτός ενωσιακού προϋπολογισμού απαιτούνται για τις διμερείς συνεργασίες. Αυτό τεκμηριώνει πόσο σημαντική είναι η συζήτηση που πρέπει να γίνει σε επίπεδο αρχών με το Συμβούλιο. Το ίδιο σημαντικό είναι το θέμα των διοικητικών επικαλύψεων. Αυτό πρέπει να το δούμε καλύτερα μαζί με το Συμβούλιο να μπει στη συζήτηση. Για τις πολιτικές προτεραιότητες έχουμε προσθέσει νέες παραγράφους εις ό,τι αφορά τη θαλάσσια πολιτική, τον τουρισμό, ως νέα καθήκοντα που προκύπτουν από τη συνθήκη και πρέπει να μας απασχολήσουν για να δούμε πώς θα αντικατοπτρίζονται αυτές στον προϋπολογισμό. Τώρα για τα δύο μεγάλα μπλοκ, χωρίς να παραγνωρίσω τα άλλα σημαντικά θέματα, έρευνα, καινοτομία, υποδομές και την σχετική χρηματοδότηση, συμπεριλαμβάνοντας και καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα και μηχανισμούς στη γεωργική πολιτική, το σύστημα των δύο πυλώνων, αυτό το υποστηρίζω ρητά, όπως και τη συμβολή της κοινή αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία. Και αυτό το καθεστώς συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης των συστημάτων θέλουμε να το επιτύχουμε για να δείξουμε στην Κομισιόν ότι πρέπει να απασχοληθεί όχι μόνο με την πράσινη γεωργία αλλά και την πολλαπλή συμμόρφωση, την αποτελεσματικότητα και να ε, είναι ε, ε, καλύτερα, να διασφαλίζεται καλύτερα η πολιτική. Σε όλους τους τομείς απαιτούνται πολλά πράγματα. Πρέπει να αποφύγουμε τις ρήξεις. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τις χώρες συνοχής όπως λέγονται, αλλά αφορά όλη την επικράτεια, όλο το έδαφος της Ένωσης. Παντού ε, θα πρέπει να αποφύγουμε ρήξεις, γιατί η προβληματική που αναφέρθηκε πριν ισχύει και για το δικό μου ομόσπονδο κρατήδιο και τη δική μου εκλογική περιφέρεια που δεν είναι χώρα συνοχής. Ε, χωρίς ε, τη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό δεν μπορούμε και εμείς να κινηθούμε όμως. Θα πρέπει επίσης να δούμε το ρόλο της ολοκλήρωσης στρατηγικής 2020. Το θέμα της συγχρηματοδότησης το θίξαμε. Ε, ε ενισχύσει στη μεταβατική περίοδο και τα προβλήματα δύσκολων περιφερειών και από δημογραφικής άποψης δύσκολες και από μακρισμένες περιφέρειες όλα αυτά τα θίξαμε. Βλέποντας όλες τις τροπολογίες νομίζω ότι είναι δυνατόν ο εισηγητής να καταλήξει σε καλές συμβιβαστικέ τροπολογίες. Καλώς. Αυτά για το πρώτο... Ναι, για το πρώτο μέρος θέλετε να μιλήσετε κι εσείς. Ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λεπτομέρειες σχετικές με την πολιτική συνοχής. Το πρώτο που θα ήθελα να πω σχετικά με το phasing out και το θέμα των δύο κατηγοριών, σύγκληση και ανταγωνιστικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την δημιουργία μιας ενδιάμεσης κατηγορίας. Σύμφωνα με τον κύριο Κλουτ, θα εμποδίζει να περνάνε απότομα οι περιφέρειες ε, από την κατηγορία σύγκλησης στην κατηγορία ανταγωνιστικότητας. Νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την ιδέα. Επιτρέπει όπως είπα να υπάρξει ένα πιο σταδιακό πέρασμα και επιτρέπει επίσης να υπάρξει και μία συνέχιση της πολιτικής συνοχής. Εφόσον δεν περιμένει βοήθεια σε σχέση με την κοινωνική συνοχή η περιφέρεια, θα πρέπει έτσι και αλλιώ να έχει σαν στόχο να αποκτήσει πραγματική ανταγωνιστικότητα. Πρέπει λοιπόν σε σχέση με αυτήν την ενδιάμεση κατηγορία να εμείνουμε για να διασφαλιστεί η συνέχεια της πολιτικής. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι με περιορισμένο προϋπολογισμό πρέπει για αυτή την πολιτική να εργαστούμε όπως έχει ήδη προταθεί για θέματα χρηματοδότησης νοτόμα. Αντί να χρηματοδοτούμε ή να συγχρηματοδοτούμε μέσω επιδοτήσεων άμεσα τις επιχειρήσεις και τους τοπικούς γενικά εμπλεκομένους, καλό θα ήταν να είχαμε δανειοδοτικά συστήματα επιδοτουμένου επιτοκίου στη διάθεσή μας, με, με διαφοροποιούμενους ρυθμούς απόσβεσης που θα επιτρέψουν ε, οι επιστροφές, ε, την χρηματοδότηση και άλλων προγραμμάτων, κάτι το οποίο δεν ισχύει με τις ε, επιδοτήσεις. Η πολιτική λοιπόν αυτή μπορεί να καταστήσει την Ευρώπη συγκεκριμένη στα μάτια των πολιτών μας. Είναι μια πολιτική που δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιπαραθέσουμε με την ΚΑΠΑ άλλωστε. Ευχαριστώ. Φτάνουμε στο τέλος της συζήτησης για το πρώτο τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να περάσουμε αμέσως στο δεύτερο τμήμα. Για το δεύτερο τμήμα λοιπόν. Τεχνικές πλευρές <clears throat> της διάρθρωσης. Και το τρίτο τμήμα θα είναι το θέμα των πόρων και το επίπεδο, το ύψος των πόρων. Λοιπόν, ο Σαλβαντόρ θέλει να κάνει κάποια παρατήρηση. Ναι, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. διότι εγώ είμαι σε χειρότερη θέση από τους συναδέλφους που πήραν το λόγο, διότι δεν έχω μπροστά, δεν είχα μέχρι τώρα τις ε, συμβαστικές τροπολογίες. Ενώ οι συνάδελφοι έχουν τις ε, τροπολογίες που καταθέσει κάτι πολιτική ομάδα. Θα πω το εξή. Μεταξύ θετικών και αρνητικών προτεραιοτήτων θα πω το εξής. Για τις θετικές υπάρχει γενικότερη συνένεση μεταξύ όλων. Δηλαδή θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις δαπάνες για πολιτικές που προσδίδουν την ε, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Πράγμα που σημαίνει ότι και στους εθνικούς προπολογισμούς θα υπάρχει οικονομία. Επίσης, η στρατηγική 2020 δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ο οδηγός. Υπάρχει συνένεση ότι αυτή η στρατηγική θα πρέπει να είναι σαφέστατη και να ξέρουμε συγκεκριμένα σε τι κονδύλια ανέρχεται για να μην αποτύχουμε όπως και με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Τώρα, μεταξύ των προτεραιοτήτων, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιοχ, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αηφόρος ανάπτυξη, συνοχή, έρευνα, ανάπτυξη, όλα αυτά τα θέματα είναι προτεραιότητες και υπάρχουν τροπολογίες των κρατών μελών για να θεσπίσουμε νέες προτεραιότητες. Η ισότητα των φύλων, κοινωνική πολιτική, νέοι, ε, ναυτιλιακή πολιτική, τουρισμός, αθλητισμός και τα λοιπά. Ο εισηγητής ούτως ή άλλως θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα αυτά τις προτάσεις όταν θα κάνω εγώ τις συμβαστικές μου τροπολογίες. Επίσης πιστεύω ότι εγώ προσπαθώ και τις διάφορες παραδοσιακές πολιτικές να τις ε, προσπίσω, δεδομένου ότι είναι αυτές που είναι οι πιο ορατές από τους πολίτες και είναι από τις προτεραιότητές μας. Θα πρέπει να τις διατηρήσουμε λοιπόν. Απ' την άλλη, όσον αφορά την ΚΑΠ, Αναφέρθηκε επίσης ότι τελικά ως ΣΟΥΡ δεν είμαστε αυτοί που θα θεσπίσουμε τα όρια της ΚΑΠ. Η πολιτική θέση είναι αν θα αποδεχθούμε ή όχι τη μεταρρύθμιση την οποία προβλέπει ο Επίτροπος Τσόλος από την Επιτροπή. Και υπάρχει σχετική έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας, άρα δεν μπορούμε να μπούμε στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Γεωργίας. Αλλά μπορούμε να ενσωματώσουμε κάποιες θεμελιώδεις ιδέες. Δηλαδή ότι η ΚΑΠ δεν θα πρέπει να λάβει μειωμένα κοινοτικά κονδύλια, αλλά απ' την άλλη θα πρέπει να βασίζεται σε κανόνες πολύ πιο αυστηρούς από ό,τι στην προηγούμενη, ε, με την προηγούμενη ε, δημοσιονομική πειθαρχία. Τώρα, θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι δυνατότητες απορρόφησης. Διότι υπάρχουν οι διαφορές μεταξύ πιστώσεων υποχρεώσεων και πληρωμών και θα πρέπει να δούμε πώς χρησιμοποιήθηκαν για να μπορέσουμε να καταλήξουμε συμπεράσματα. Να δούμε πώς ανταποκρίθηκαν τα κράτη-μέλη, πώς μπορούσαν να απορροφήσουν τα κράτη-μέλη τις διάφορες πιστώσεις για την συνοχή που τους χορηγούσε ο κοινοτικός προπολογισμός. Επίσης, έγινε λόγος για ένα αντικειμενικό στόχο μεταβατικό. Εγώ την ε, ιδέα θα τη μελετήσω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να πούμε σε λεπτομέρεια στην ΣΟΥΡ, διότι η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής τη στιγμή που θα πρέπει να εκπονήσει τους κανονισμούς για την πολιτική συνοχή να το κάνει αυτό. Θα πρέπει λοιπόν όταν μιλούμε για, επειδή υπάρχουν λοιπόν στην ενοχή, θα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες όταν μπούμε στις λεπτομέρειες του προϋπολογισμού και η συνοχή θα πρέπει να συμμετάσχει και στην υλοποίηση των στόχων του στρατηγικής του 2020. Τώρα, οι αρνητικές ε, προτεραιότητες. Εγώ ως ηγητής δεν μπορώ στις παραδοσιακές πολιτικές να, δω, να πω ποιες είναι οι αρνητικές. Όχι ότι δεν θα υπάρχει συνένεση και είναι και άδικο οι γεωργοί, οι Ευρωπαίοι να πληρώσουν τίμημα για να μπορέσει να δοθεί νέα όθηση μικρομεσαίας επιχειρήσης. Θα ήταν άδικο για τις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης να χρειαστεί να συνεισφέρουν για την ε, ανάπτυξη αποδοτικών μορφών ενέργειας. Πού έχουμε αρνητικές ε, προτεραιότητες στην κατηγορία 5, στη διοίκηση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί κατά την α τρόπο να το εκθέσουμε. Αλλά ε, οποιαδήποτε πολιτική υπερψηφίσουμε εδώ ή στο Κοινοβούλιο θα πρέπει όντως να προτείνουμε περικοπή όχι στα λειτουργικές δαπάνες αλλά στις διοικητικές. Ίσως λίγο κάτω του επίπεδου προπολογισμού, ίσως με κάποιες προτάσεις ε, για τα κτίρια, για κάπου αλλού που θα μπορούσαμε να κάνουμε οικονομίες, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι το γενικό στα αρνητικά, απλώς να επικεντρωθούμε περισσότερο στις διοικητικές δαπάνες στην ε, κατηγορία 5. Μάλιστα. Κλείνουμε το πρώτο μέρος λοιπόν. Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι όταν καθορίζουμε πολιτικές προτεραιότητες χρειαζόμαστε και ανθρώπους που θα επεξεργαστούν αυτές τις πολιτικές που θέλουμε εμείς να εφαρμοστούν. Η συζήτηση αυτή θα γίνει στις 9 Μαΐου και ελπίζω ο αρμόδιος επίτροπος να μπορέσει να παρευρεθεί. Αυτό θα το μάθουμε την επόμενη εβδομάδα. Και τότε θα ξανασυζητήσουμε το θέμα της διοίκησης. Αυτό που είπε ο Κάρλ για την κατάργηση ε, της, ε, και μια έδρα συγκέντρωση όλων των, μηχανισμών, των οργανισμών στις Βρυξέλλες. Όλα αυτά θα ήταν διοικητική ελάφρυνση και από άποψη δημοσιονομική. Το ερώτημα είναι θα τα γράψουμε εμείς όλα αυτά. Ή θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ή να μην αποφανθούμε. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος, δομή, τεχνικά θέματα. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε γύρω με τις πολιτικές ομάδες. Ποιος ζητεί το λόγο. Άιμα και μετά ο Ράιμαρ. Ευχαριστώ για τις σε Ένα σχόλιο προς τον Σαλβαδόρ. Να μην ξεχνάμε ότι οι λεγόμενες αρνητικές προτεραιότητες δεν είναι θέμα αξιολόγησης μεταξύ τους ε, ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτικές, αλλά αξιολογήσεις στο εσωτερικό των πολιτικών στο εσωτερικό της κοινή αγροτικής πολιτικής κάποια θέματα δεν θα τα απρασπιστούμε όπως οι επιδοτήσεις στις εξαγωγές. Αλλά υπάρχουν άλλα τα οποία θα στηρίξουμε. Μιλάμε για ένα δύσπερι που στην κοινή αγροτική πολιτική, πολύ σοβαρά ποσά και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάζουμε τις πολιτικές στο εσωτερικό τους, στο περιεχόμενό τους και όχι να συγκρίνουμε μόνο διαφορετικές πολιτικές για τη διάρθρωση. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ισορροπήσουμε την ανάγκη για διαφάνεια, σωστή παρουσίαση, ενημέρωση των πολιτών, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν, οι πολιτικοί, οι εθνικοί πρέπει να γνωρίζουν τι δαπανούμε στον τομέα της ενέργειας, τι δαπανούμε στη γεωργία και απαιτείται φυσικά όλα αυτά να κατανεμηθούν σωστά και να υπάρχει ε, ενημέρωση για αυτά. Δημιουργούνται όμως προβλήματα στην ευελιξία όταν υπάρχουν κάτω από ένα τίτλο ε, πολύ μικρότερα, ε, ε, πολύ μεγάλη κατάτμιση. Αν υπάρχει ευελιξία μπορούμε να έχουμε πάρα πολλούς τίτλους βέβαια για να αυξήσουμε την ορατότητα αν θέλετε. Αλλά αν δεν υπάρχουν κανόνες για την ευελιξία πρέπει να είμαστε πολύ ευέλικτοι και πολύ ευαίσθητοι σε σχέση με την δημιουργία υπερβολικά μεγάλου αριθμού λεπτομεριακών αναφορών. Συνδέεται λοιπόν το θέμα με τη συζήτηση για την ευελιξία. Πρέπει να υπάρξει μια από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Παρουσιάσαμε μια τροπολογία η οποία λέγει ότι εμείς θέλουμε τρεις τίτλους, ένα για τα εσωτερικά, ένα για τα εξωτερικά και ένα για τη διοίκηση. Ιδιαίτερα στα θέματα των εσωτερικών πολιτικών χρειάζεται να υπάρξουν κάποια υποθέματα και εγώ προτείνω τέσσερα. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Είμαστε διατεθειμένοι να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά σε σχέση με την ευελιξία. Να σας ενημερώσω λέγοντας ότι στο εσωτερικό της πολιτικής μας ομάδας έγινε μια πάρα πολύ έντονη και ενδιαφέρουσα συζήτηση για το αν θα υπάρξει ξεχωριστός τίτλος για τα πολύ μεγάλα προγράμματα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. να ξεχωριστούν από τα υπόλοιπα τα πολύ μεγάλα αυτά προγράμματα, χωρίς όμως να φίξουμε τις άλλες προτεραιότητες. Το θέμα που τίθεται είναι, εμείς αυτή τη στιγμή προστατεύουμε τα μεγάλα προγράμματα ή τα μικρά προγράμματα. Εδώ υπάρχει ε, μια, ένας δισταγμός ένα θέμα σαν το ίτερ σαν παράδειγμα δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο άλλες, ε, άλλα προγράμματα στα πλαίσια του εβδόμου προγράμματος. Λοιπόν τώρα για τη διάρκεια. Έχει ενδιαφέρον να βλέπει κανείς τις διάφορες τροπολογίες. Υπάρχει μια τάση στις περισσότερες πολιτικές ομάδες ταύτισης, ευθυγράμμισης της διάρκειας ε, ε, σε επίπεδο αρχής με τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής εντολής. Το θέμα είναι μπορούμε να το κάνουμε τώρα, μπορούμε να έχουμε μια απλά πενταετή περίοδο ή θα πρέπει να υπάρχει μια πενταετής περίοδος συν. Εμείς είμαστε υπέρ της ευθυγράμμισης της διάρκειας αυτής ε, με την κοινοβουλευτική εντολή, αλλά νομίζω ότι τελικά ίσως να χρειάζεται μια επταετής περίοδος έτσι ώστε να προλάβουμε την επόμενη εντολή. Ένας από τους λόγους είναι ότι δεν είμαι βέβαιος ότι το 7 χρόνια είναι σωστό, ίσως να χρειαστούμε και 8 χρόνια. Γιατί αλλιώς ο χρόνος διαπραγμάτευσης για τη νέα Επιτροπή και το νέο Κοινοβούλιο το 2019 θα είναι πάρα πολύ μικρός και δεν θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε το πλαίσιο για μετά το 2020. Κάτι για το οποίο είμαι βέβαιος πάντως είναι ότι αν πράγματι υπάρξει μια επταετής εντολή, είτε από τώρα είτε για τώρα είτε για πάντα, ή αν έχουμε μία περίοδο άνω των 5 ετών, εν πάση περιπτώσει, 5 συν 5 κτλ. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε νομικά δεσμευτικά ε, την αναθεώρηση ανά πενταετία. Είναι, θα έλεγα, απόλυτος σε αυτό. Δεν μπορεί το Συμβούλιο να μην δεχθεί αυτή την πενταετία αναθεώρηση, εφόσον ξεπερνάμε τα 5 χρόνια. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν μια ρύθμιση 5 συν 5, αλλά οι αριθμοί και οι δείκτες για το δεύτερο τμήμα της περίοδου αυτούς θα είναι ενδεικτικοί θα έλεγα μόνο. Θα πρέπει να υπάρχει μια ενδιάμεση αναθεώρηση, κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι πλήρως υποχρεωτικό. Ευχαριστώ Ράιμερ και μετά η Χέλγα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα βρούμε τελικά κοινή λύση. Σύμφωνο με τον Γκέραν, η δομή, η διάρθρωση είναι σημαντική για την ορατότητα ο εισηγητής προσπάθησε να επιτύχει ένα μείγμα μεταξύ της ολοκλήρωσης ε, της στρατηγικής 2020 και των άλλων τομέων που δύσκολα εντάσσονται, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απλό να ενταχθεί η Ευρώπη 2020 στα πλαίσια της ανάπτυξης χωρίς, αποκλεισμού, ε, χωρίς αποκλεισμούς, ανταγωνιστική, βιώσιμη κλπ. Καλό είναι λοιπόν να εξετάσουμε το θέμα. Η ομάδα μας κατά πλειοψηφία έκανε πρόταση να ε, καταθέσουμε τροπολογίες και σε ό,τι αφορά τη σειρά και στην sustainable development, ε, μεταφορές, ενεργειακές πολιτικές, ε, αυτά να είναι σε χωριστό υποκεφάλαιο και με τη σειρά να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα και την επισητιστική ασφάλεια. Με βάση την εμπειρία από τη δομή μέχρι τώρα και επειδή πιστεύουμε ότι καλύτερα θα συντεριάζονται έτσι οι επιμέρους τομείς. Γνωρίζω ότι υπάρχουν τροπολογίες από την ομάδα μου που προτείνουν το 1β και το 1γ να τα συγχωνεύσουμε, αλλά αυτά θα τα δούμε όλοι μαζί, ανεξάρτητα από το θέμα της δομής ε, που θα συζητηθεί. Η συνθήκη προβλέπει λιγότερες κατηγορίες, πρώτον και δεύτερον, έχει δίκιο ο Γκέραν, δεν πρόκειται για το αν θα έχουμε τρεις ή πέντε ή έξι κατηγορίες, το σημαντικό είναι τι κανόνες θα τα διέπουν όλα αυτά, πώς θα δεσμευθούμε, τι συμφωνίες θα υπάρχουν για να υπάρχουν τα κατάλληλα περιθώρια ή ευελιξίες για τους διάφορους τομείς πολιτικής. Δεν θα πρέπει δηλαδή οι ε, κατηγορίες να μας κάνουν ε, λιγότερο ευέλικτους και να μας μπετονάρουν τις πολιτικές. Εκτός αυτού σκεφτήκαμε και μια πρόσθετη συμπληρωματική κατηγορία για δαπάνες εκτός του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ε, για να καταγράψουμε αυτά που διοργανώνονται εκτός προϋπολογισμού και να έχουμε μια γενικότερη εικόνα. Νομίζω ότι πρέπει και το Κοινοβούλιο και για την ε, ενότητα του προϋπολογισμού να κάνει αυτή τη συζήτηση με το Συμβούλιο. Τώρα, η προστασία, το ring fencing των μεγάλων έργων, ως σκέψη εξετάστηκε και από εμάς και μας βρίσκει σύμφωνους γιατί βλέπουμε αυτή την προβληματική. Από τη μια αρνείται το Συμβούλιο τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Σιγά σιγά εγκρίνονται οι περαιτέρω χρηματοδοτήσεις ε, και παράλληλα έτσι έχουμε το μόνιμο πρόβλημα της αναδιάρθρωσης του προϋπολογισμού. Για να έχουμε σαφέστερη προοπτική, πρώτα να μιλήσουμε για τα ε, έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό ως μεγάλα έργα, τι θα στοιχήσουν και πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου δεν θα υπονομευθούν και παραμεριστούν. Αν δεν διασφαλίζονται αυτά στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό πρέπει να δούμε ποια έργα είναι σωστά και ποια δεν είναι και να συζητήσουμε τότε και τις αρνητικές προτεραιότητες. Υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να περιγράψουμε τι ακριβώς εννοούμε. Μετά το θέμα των, της ευελιξίας έχει συζητηθεί πολλές φορές. Νομίζω ότι η νομοθετική ευελιξία όπως υφίσταται σήμερα είναι αρκετή, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ποτέ δεν την αξιοποιήσαμε 100%. Μιλήσαμε για 7-10% νομοθετική ευελιξία. Μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο μας με αυτό. Τώρα, τα περιθώρια που δεν έχουν αξιοποιηθεί θα πρέπει να αξιοποιηθούν περισσότερο. Αλλιώς δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο πολιετές. Ε, τώρα, για τα χρονοδιαγράμματα. Η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ε, τίνει να συμφωνήσει στα 7 χρόνια, όχι γιατί αυτό είναι θέμα συνταγματικό, συνταγματικής νομιμότητας, αλλά γιατί απλοποιεί την δομή και τη λειτουργία των προγραμμάτων που υπάρχουν στο πολιετές πλαίσιο. Ακόμη δεν έχουμε βρει μία ε, απλουστευμένη διαδικασία. Καλό είναι λοιπόν σε αυτό το στάδιο να δεχτούμε την επταετία χωρίς να αποκλείουμε και τα πέντε χρόνια. Στην τελευταία φορά που συνεδριάσαμε, ακριβώς σε αυτό το θέμα, ε, είχαμε μια σχετική διατύπωση και στα ψηφίσματα η μένα ανάφεραν τα πέντε χρόνια, οι άλλοι τα επτά. Μπορούμε λοιπόν εδώ να ρίξουμε γέφυρες, να μην αποκλείσουμε τα πέντε χρόνια. Μπορούμε να δούμε τις σχετικές τροπολογίες που δεν είναι από την ομάδα μας για ειδικά έργα μπορούμε να έχουμε πολιτικές συμφωνίες που θα υπερβαίνουν την πενταετία. Αυτό μπορεί να αποτελεί μέρος μιας συμβιβαστικής λύσης. Εν τω μεταξύ, με βάση την πείρα που αποκομίσαμε από τις υποχρεώσεις μας, το 5 συν 5 μπορεί να ισχύσει όταν, είναι, όταν υπάρχουν νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις του Συμβουλίου. Αυτά όμως θα μεταφραστούν σε πραγματικότητα. Ίσως ε, θα πρέπει να τροποποιήσουμε τη συμφωνία μας ε, και εκεί ανησυχώ λίγο ε, με βάση την εμπειρία του παρελθόντος ε, αν ταχθούμε υπέρ της επταετίας χωρίς να αποκλείω άλλα, αυτό είναι μια καλή λύση για να διασφαλίσει και το Κοινοβούλιο τα συμφέροντά του. Αυτό σημαίνει σε τελευταία ανάλυση ότι πρέπει να συμφωνήσουμε για μια αλλαγή. Και πραγματικά εδώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο Συμβούλιο. Helga, jetzt, bitte. Ja, vielen Dank, Jutta. Helga, ευχαριστώ Γιούτα. Καταρχήν η Επιτροπή μας, η Ειδική Επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής. Προκλήσεις τι επίκειται, πού πρέπει να αντιδράσουμε, τι νέα προβλήματα υπάρχουν και τι μεγάλα ζητήματα πρέπει να μας απασχολήσουν μέχρι το 2020. Και δημοσιονομική πόρη για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση. αυτό είναι ο τίτλος της ειδική Επιτροπής. Όλα αυτά κρύβουν ένα πολιτικό νόημα, υποθέτω. Πρέπει λοιπόν από κοινού να αναρωτηθούμε τον τίτλο αυτόν πώς μπορούμε να τον δικαιώσουμε με βάση την έκθεση αυτή. Πρέπει να πω στον Σαλβαντόρ ότι επιμένουμε πολύ στα παλιά πράγματα, στις παλιές καταστάσεις. Παραδείγματα, όταν μιλάμε για προκλήσεις και για τη βιωσιμότητα, ε, επιδοτούμε την καλλιέργεια καπνών. Τα τελευταία χρόνια είχαμε τις εξαγωγικές επιδοτήσεις. Στην πολιτική αλληλείας η Κομισιόν η ίδια διαπιστώνει ότι δεν είναι βιώσιμη, αλλά έχει αποτύχει. Όμως εμείς μιλάμε για βιώσιμη Ευρω... Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με τον Γκέραν ότι δεν είναι δυνατόν όταν μιλάμε για αρνητικές προτεραιότητες να μιλάμε μόνο για διοικητικές δαπάνες. Σωστό και αυτό, να το δούμε. Αλλά εμείς θέλουμε να μιλήσουμε, φιλοδοξούμε να μιλήσουμε για τις μεγάλες προκλήσεις και αυτό πρέπει να γίνει σε όλους τους τομείς πολιτικών μας. Δεν μπορούμε να διαπιστώνουμε ότι στην ε, πολιτική συνοχή ή στην ΚΑΠ θα πρέπει να παραμείνουμε στα παλιά. Αυτό δεν συνάδει με το στρατηγικό ερώτημα ε, σχετικά με τις σύγχρονες προκλήσεις και τι πρέπει να κάνει τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εσωτερική πολιτική, την ενιαία πολιτική. Μιλάμε για εξυγίανση. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τη, τα διαρθωτικά ταμεία, πρέπει να αξιοποιήσουμε την γεωργική πολιτική. Αλλά η Επιτροπή μας θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τις ε, αρμόδιες επιτροπές, αλλά η έντολή μας περιλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής προτάσεων. Αυτό είναι το καθήκον μας και δεν πρέπει να το αμελήσουμε. Αλλιώς δεν θα έχουμε ανταποκριθεί στο έργο που αναλάβαμε. Γι' αυτό προσπαθήσαμε και οι πράσινοι να κάνουμε κάποιες προτάσεις και για τους τίτλους, τι πρέπει να αλλάξει να μην κρατήσουμε μόνο τα παλιά, αλλά με τεκμηριωμένο τρόπο να πούμε ποιο μπορεί να είναι ένα καλύτερο μοντέλο και πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε πλειοψηφίε υπέρ αυτού του νέου μοντέλου. Κάναμε και μία πρόταση για ένα χωριστό κεφάλαιο για την ευελιξία και για τα μεγάλα έργα υποδομών. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνηγορούν υπέρ μιας τέτοιας προσέγγισης. Έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε έμφαση ε, σε άλλους τομείς πολιτικής και να συμφωνήσουμε. Ξέρω από τη χώρα μου και από την Υπουργό Γεωργίας ότι πολλές φορές δεν είμαστε στο ύψος της νέας εποχής και των νέων προκλήσεων. Άρα λοιπόν εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να μείνουμε στα παλιά γνωστά συστήματα αλλά να ανταποκριθούμε στο καθήκον που αναλάβαμε από το Κοινοβούλιο να είμαστε σοβαροί και να δείξουμε προθυμία αλλαγών με αφετηρία τους στόχου που από κοινού αποφασίσαμε. Περισσότερη σοβαρότητα λοιπόν και κινητικότητα γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα καθήκοντα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Τώρα, όταν θα δώσω το λόγο στους επόμενους ομιλητές, θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι που ενδεχομένως ξεχάσαμε, Χέλγα, ότι είμαστε στο σημείο 2 των τροπολογιών, στο μέρος 2, δηλαδή δομή, διάρθρωση και τεχνικά θέματα, η Κωνσταντσε. Ναι, αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε μια σύντομη παρατήρηση. Κυρία Τρούπελ, διαβάστε την έκθεση Καρίγκα, το εδάφιο για την ε, πολιτική συνοχής. Θα πρέπει να το καταλάβουμε. Όταν μιλήσουμε για αλλαγή κλίματος, έρευνα, ανάπτυξη και όταν λέμε ότι αυτά είναι κύριες προτεραιότητες στην πολιτική συνοχής, μιλάμε για εξυγχρονισμό της πολιτικής συνοχής. Αν ευπροηγουμένο εξυγχρονισμό, Τι άλλο θέλετε. Αφήστε μας να δουλέψουμε αυτούς τους τομείς και μην ζητάτε συνεχώς καινούργια πράγματα για να ακούγεστε ωραίοι και αρεστοί. Νομίζω ότι μπήκαμε σε μια τροχιά και πρέπει να τη συνεχίσουμε. Σε αυτά τα πλαίσια θέλω να υπενθυμίσω ε, σε όλους τους συναδέλφους ότι είμαστε κεφάλαιο 2 και εδώ είμαστε βέβαια, αλλά όχι μόνο, αλλά ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα μηχανισμός, ένα μέσον. Θυμάστε τι ε, έγραψε ο Γιάνν Όλμπριχ για το μέσο αυτό. Τι θα, θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα το μέσον. Μην ανακατεύουμε όμως την νομοθεσία. Εντάξει. Ο Ρίτσαρντ Έλσουρθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα, για την διάρκεια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Νομίζω ότι είναι θέμα ισορροπίας. Καταλαβαίνω τα τεχνικά επιχειρήματα. Δηλαδή, αν κάνει κανείς μακροπρόθεσμες επενδύσεις, καλύτερα να έχει και έναν ε, ανάλογο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. Για να πιο Θα πρέπει όμως να βρούμε την ισορροπία. Και θα πρέπει να υπάρχει και η πολιτική αξιοπιστία, η λογοδοσία εκ μέρους ημών. Διότι Όσον βλέπω, αυτό είναι κάτι το οποίο λείπει αυτή τη Εάν λοιπόν η διάρκεια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου ε, ε μπορέσει να εξωθεί με τις... Ε, ε, uh, είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε πολύ πιο πολιτικό το όλο θέμα. Και κατά την άποψή μου αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι θετικό. Τώρα, όσον αφορά τα διάφορα κεφάλαια, εγώ είμαι ανοιχτό, αλλά νομίζω ότι και πάλι είναι θέμα ισορροπία. Κατανοώ απόλυτα ότι θέλουμε να έχουμε ευελιξία στον προπολογισμό και όντω αν ε, είμαι από αυτού που είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάπου πάγωμα, νομίζω ότι μπορώ να πω εξίσου ότι η ευελιξία είναι επίση σημαντική. Θα πρέπει όμως να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ασκήσουμε και τον ε, έλεγχο και την ε, δημοσιονομική ε, πειθαρχία. Για προγράμματα όπως το Γαλλίο και άλλα, δεν είναι ότι διαφωνώ, αλλά δεν συμφώνησα με τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτήθηκαν και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο έλεγχος. Και πάλι λοιπόν νομίζω ότι εδώ κάτι θα πρέπει να συζητήσουμε. Αυτά θα συζητήσουμε μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Θα ήθελα να επανέλθω στις ε, πρωτοβουλίες, Πρόεδρε. Διότι ήθελα να πω σε σχέση με την ΚΑΠ και τη χρηματοδότησή της, ακούγοντα τα προσεγητής για τις υποχρεώσεις της συνθήκης, ότι εκεί αναφέρονται ε, θέματα τα οποία αφορούν τον πρώτο πυλόν τη κόπας. Στον πυλώνα 2 υπάρχει θέματα περιφερειακά, υπάρχουν ε, άλλα θέματα τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά από συνθήκες, άρα Μπορούμε να τα συζητήσουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο τα κάνουμε όλα αυτά. Και εσεί ε, ζητήσατε να υπάρχει μεγαλύτερη κουρικότητα εδώ. Εγώ ζητώ συγχρηματοδότηση ώστε να μπορέσουμε όταν υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, κάποια κενά να τα συμπληρώσουμε. Αλλά θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα ε, υποχρεώσεις ε, ε, στον πρώτο πυλώνα για την ΚΑΠ δεν αναφέρονται σε θέματα του αγωνιστικότητας. Ευχαριστώ. και μετά η Σοφή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λίγα σχόλια σύντομα. Πρώτον, έχουν προταθεί πολλές επιλογές για την αρχιτεκτονική της πρότασης και για το ποια θα πρέπει να είναι η δομή τελικά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε λίγους τίτλους και πρέπει το σύνολο των πολιτικών να τα εντάξουμε σε ένα κεφάλαιο. Όλοι θέλουμε την ευελιξία. Ξέρουμε όμως ότι για να το πετύχουμε χρειάζονται όσο λιγότερα κεφάλαια ε, είναι απαραίτητο τόσο το καλύτερο για την οικονομική διακυβέρνηση. Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφερθούμε στο θέμα αυτό, δεν ξέρω τι θα βάλουμε μέσα σε αυτό. Όλα αυτά τα προγράμματα, οι μηχανισμοί σταθεροποίησης κτλ. χρηματοδοτούνται περισσότερο όχι από τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά από τα κράτη-μέλη. Για τη διάρκεια επίσης. Θα υποστηρίξω ότι τα 7 χρόνια θα πρέπει να μείνουν μέχρι το 2020 και μετά ίσως να χρειαστεί να περάσουμε στη λογική του 5 συν 5. Αλλά εφόσον είμαστε βέβαιοι βέβαια ότι υπάρχει η νομική βάση για να το πετύχουμε αυτό. Δεν απαιτείται μόνο μία νομική βάση για να διασφαλίσουμε την συνέχιση των προγραμμάτων, αλλά θα πρέπει στα πλαίσια της ενδιάμεσης ε, αναθεώρησης, η οποία πρέπει να είναι απαραίτητη, να συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Ευχαριστώ πολύ, Σοφή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την ε, δομή του προπολογισμού. Εγώ κατέθεσα τροπολογίες για το κεφάλαιο αυτό για μια δραστηριότητα που μου φαίνεται ότι είναι σημαντική, που είναι ο αθλητισμός, που θεωρούμε πολλές φορές ως κάτι το δευτερεύουσα σημασία. Πρόκειται όμως για μια οικονομική δραστηριότητα και θα σας πω ότι αυτή η δραστηριότητα στην Ευρώπη χρειάζεται έλεγχο κανονισμούς, εναρμόνιση και στο δημόσιο τομέα και για κάποιες ε, χρηματοπιστωτικές και οικονομικές δραστηριότητες. Είμαι, φεύγω εκτός προπολισμού, νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι ο αθλητισμός σίγουρα θα δώσει και κάποια νέα πνοή στις πολιτικές μας σε σχέση με τον τρόπο προσεγγίλουμε τους πολίτες. Είμαι στη διάθεση του εισηγητή, διότι πιστεύω ότι δίνει νέα ψυχή στην Ευρώπη ο αθλητισμός και πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για τα διαρθρωτικά και τον προϋπολογισμό. Σημαντικό είναι να δούμε τη διάρκεια. Δεν έχουμε θέση ως κοινοβούλιο, άρα αν δεν πάρουμε θέση δεν έχουμε πιθανότητες απέναντι στο Συμβούλιο. 7-8 χρόνια κάτι πρέπει να αποφασίσουμε. Τι θέλουμε. Εγώ νομίζω ότι ο πιο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός πάνω από 5 χρόνια δεν έχει νόημα μεγάλο θεωρώ λόγω των ταχυτάτων αλλαγών αναδιαρθρώσεων. Δύσκολο να βάλουμε ένα πλαίσιο. Ε, πολλοί είπαν να μείνουμε στο, στα 7 χρόνια στον προϋπολογισμό του 11, στα γεωργικά έχουμε 1,6 δις περιθώριο. Άγνωστο πόσα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν στο τέλος, καθοριστικό όμως ότι στα πλαίσια που αναφέραμε θα υπάρξει αλλαγή μεγάλη στις βιομηχανικές περιοχές και θα υπάρξουν και κλασικές διαρθρωτικές αλλαγές στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν και δημοσιονομικά πρέπει να μπορούμε να αντιδρούμε. Μπορεί σε κάποιους τομείς να χρειαστούν περισσότερες επενδύσεις από ό,τι σε άλλους είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια πανευρωπαϊκή συζήτηση. Αυτό το θέλουν οι συνάδελφοι πράσινοι, για να μιλήσουμε για τα πυρηνικά. Αλλά αν μιλήσουμε σε αυτό το επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι και από τον προϋπολογισμό να αντιδρούμε. Να επενδύουμε περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη, να η φόρο ανάπτυξη βιώσιμη κλπ. Άρα Δύο πράγματα πρέπει να ρυθμίσουμε στον προϋπολογισμό και στην έκθεσή μας. Πρώτον, διάρκεια του πλαισίου, δημοσιονομικού πλαισίου. Εγώ νομίζω ότι καλό είναι να μην, είμαστε, να μην είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε σχεδιασμό που θα ξεπερνάει τα 7 χρόνια. Και θα πρέπει να έχουμε και ευελιξία όσο γίνεται μεγαλύτερη, ούτω ώστε να αντιδρούμε σε οικονομικές αλλαγές ή και σε φυσικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε κάποια κράτη-μέλη όπως έχουμε δει. Σε αυτούς τους δύο τομείς να επικεντρωθούμε και εκεί να προσπαθήσουμε να πετύχουμε συνένεση. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Δεν έχω άλλους στον κατάλογο για την δομή και τη διάρκεια. Σαλβαντόρ, για να κλείσουμε το αυτό. Αρχίζω με την ευελιξία που κατά την άποψή μου στην πρώτη ανάλυση είναι το πιο απλό θέμα. Μίλησαν για αυτό το θέμα οι πολιτικές ομάδες και νομίζω ότι η παράγραφος, στην παράγραφο για την ευελιξία υπάρχει συνένεση μεταξύ ημών και ημών. Όλοι μιλάνε για την αναθεώρηση των διαφορών κατηγοριών δαπανών. Κάποιες ομάδες μιλούν περιθώριο ευελιξίας με συγκεκριμένο ποσοστό. Άλλοι ζητούν νέα ε, εργαλεία εντός εκτός του προπολισμού για την ευελιξία και πιστεύω ότι η συνένεση που υπάρχει στην έκθεσή μου για το θέμα αυτό αποδεικνύει ότι όλα ήταν σωστά στις επιλογές μου σε σχέση με τις επιδημίες των συναδέλφων. Τώρα, θα αφορά την δομή, θα το αφήσω στο τέλος. Η διάρκεια τώρα. Η διάρκεια είναι ένα θέμα που εξετάσαμε βλέποντας όλες τις δυνατότητες. Όπως ξέρετε υπήρχε μία αρχική πρόταση από το προηγούμενο Κοινοβούλιο για πέντε χρόνια για την προσαρμογή της εντολής του Κοινοβουλίου με αυτό της Επιτροπής και τις δημοσιονομικές προοπτικές. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι συγκεκριμένα για το επιχείρημα που ε, εξέφρασε ο Άλβαρο, εγώ θα χρησιμοποιήσω το αντίθετο επιχείρημα. Συγκεκριμένα τη στιγμή που υπάρχει πολύ λίγη ασφάλεια για το σφαιρικό οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια, είναι καλό, κατά την άποψή μου, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να είναι το πιο σταθερό δυνατό. Και αυτό σημαίνει 7 χρόνια. Βεβαίω υπάρχουν ε, μειονεκτήματα, τα γνωρίζουμε όλοι, αλλά αυτή τη στιγμή που είμαστε σε μία κατάσταση τι, όσον αφορά την ευρωπαϊκή οικονομία, νομίζω ότι η καλύτερη δυνατή πρόταση είναι διάρκεια 7 ετών. Δεν είμαι υπέρ του 5 συν 5, δεν το εμπιστεύομαι. Αυτό είναι γιατί δεν το εμπιστεύεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φαντάζομαι, διότι έχουμε και την ε, πρόσφατη εμπειρία του Συμβουλίου για τις ρήτρε αναθεώρησης μέσω πρόθεσμα. Δεν υπάρχει για αυτές τις ρήτρε ε, αρκετή συνένεση, άρα το 5 συν 5 μας κάνει 10 χρόνια και κατά την άποψή μου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ε, αυτή η χρονική διάρκεια των 10 ετών. Άρα επιμείνω στα 7 χρόνια που βλέπω ότι κατά κάποιον τρόπο καμία πολιτική ομάδα δεν απορρίπτει ρήτα. Τώρα, όσον αφορά την δομή. Το θέμα της δομής είναι πολύπλοκο, διότι κατανοώ ότι χωρίς να επηρεάσουμε την κατανομή των δαπανών, είναι σημαντικό να δούμε πώς θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε διάφορες κατηγορίες δαπανών, διότι τελικά αυτό είναι το πιο ορατό μέρος της έκθεσης δεν θέλω να έχετε την εντύπωση ότι οι θέσει των πολιτικών ομάδων είναι τόσο πολύ απομακρυσμένε ή μεν από τους δε. Ούτε η δική μου, ούτε των σοσιαλιστών, ούτε των πρασίνων, ούτε του ΕΛΚ, ούτε των φιλελευθέρων. Τώρα, για τις μικρότερες ομάδες θα πρέπει να δω ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις εδώ. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών κατηγοριών που θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά εδώ υπάρχουν και κάποια προβλήματα ορισμού. Ο εισηγητή και πρόβληση πέντε κατηγορίες, εδώ ζητούνται έξι. Έχουμε γενική συνένεση για τη συμπερίληψη της στρατηγικής 2020 ή ειδικά ως στρατηγική 2020 ή μέσω των διαφόρων συνιστοσών της, δηλαδή αηφόρος ανάπτυξη, ευφύησα και ε, συμπεριληπτική ανάπτυξη. Υπάρχουν ε, κάποιες διαφορές για την ε, συμπερίληψη ή όχι της έννοιας της δαγένειας. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερα εδώ να μιλήσουν για τις πολιτικές που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και αυτόν το αφήσουμε κατά μέρος και υπάρχει εκ μέρους των Πρασίνων μια ενδιαφέρουσα πρόταση για τη συμπερίληψη μιας ειδική κατηγορίας για το ε, αποδεματικό, πρώτα απ' όλα για την οικονομική διακυβέρνηση και το ΕΛΚ προτείνει οι δαπάνε Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιουργούνται εκτός κοινοτικού προπολογισμού επίσης να συμπεριληφθεί. Αυτό θα είναι ένα αρκετά πολύπλοκο μέρο για να μπορέσει να ευρεθεί ένα συμβαστική πρόταση που θα είναι αρεστή σε όλου. Αλλά και η Γραμματεία και εγώ κατά τη διάρκεια αυτών των επόμενων δύο εβδομάδων θα προσπαθήσουμε παρουσιάσουμε μία δομή που ε, θα ικανοποιήσει σχετικά του συναδέλφους για να το εγκρίνουν. Τελειώνοντας, ε, θα πω το εξής. Για την... Ε, ο στόχος, ποιος είναι ο στόχος του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου μεταξύ όλων και της νέας πολιτικές. Να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης και δεν θα πρέπει ένα μέρος του πληθυσμού να πληρώνει για τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Το λέω αυτό και για τη συνοχή και για την ΚΑΠ, στις οποίες θα πρέπει να γίνουν πολύ σημαντικές αλλαγές, διότι τελικά αυτό το οποίο θα πρέπει να προστατεύσουμε είναι η ευημερία και η απασχόληση για όλους τους πολίτες. Ή για τους καπνεργάτες, ή για τους επιχειρηματίες, ή για τους γεωργούς, συγγνώμη, για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία και τους επιχειρηματίες, λέει ο εισηγητής, ώστε να μην ζημιώσουμε κανένα τομέα της οικονομίας. Τώρα, με συγχωρείτε, τα μεγάλα σχέδια. Τα μεγάλα σχέδια που είναι ένα θέμα που κατατέθηκε ως εναλλακτική λύση. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Στα πλαίσια αυτής της δομής μπορώ να τα συμπεριλάβω αυτά. Αλλά βεβαίως μας λέει η πείρα ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και στον, ε, χρηματο, δημοσιονομικές ε, προοπτικές τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω πώς μπορώ εγώ αυτό να το εισαγάγω στην δομή, αλλά θα ζητήσω την βοήθεια των, και τη συνδρομή των συντονιστών. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση και στο δεύτερο μέρος και περνάμε στο τρίτο. δύο ομιλητές, αν Λουκτεάν και η Διαγκάρτια Σαμπάλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν έχει καταθέσει πολλές τροπολογίες σε σχέση με αυτό το τμήμα το οποίο μας φαίνεται αρκετά ισορροπημένο έτσι όπως είναι τα πράγματα. Όταν παρουσιάσει την τελική της πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δούμε πώς θα πάει η συζήτηση, ιδιαίτερα σε σχέση με την χρηματοδότηση. Μια συζήτηση η οποία νομίζω ότι θα γίνει με κάπως πιο έντονο τρόπο. Αυτό που έχει σημασία σε εμά είναι να ενισχύσουμε το κείμενο σε επίπεδο ασφάλειας. Θέλουμε, ε, Θέλουμε να γίνει το κείμενο πιο διαφανές και θέλουμε κατά τη διάρκεια του προϋπολογισμού να υπάρξει σαφέστατη αναφορά στο θέμα των ιδίων πόρων. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά το σύνολο των προϋπολογισμών. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το θέμα των πόρων και πρέπει να τεθεί επιτέλους το θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει το ρόλο ε, τον οποίο του δίδει η συνθήκη και η συνθήκη προβλέπει ακριβώς τη δυνατότητα παρέμβασής μας. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της διαφάνειας. Πρέπει να υπάρξουν περισσότερες εγγυήσει ε, για διαφάνεια στον προϋπολογισμό και οι εσωτερικές μεταφορές είναι κάτι το οποίο δεν καλύπτεται, θα έλεγα, πλήρως σε επίπεδο διαφάνειας. Καταθέσαμε και κάποιες τροπολογίες οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν προκλητικές. Αν παραμείνουμε στο πάγωμα των πόρων, έτσι όπως είναι, των εσόδων, τότε το Συμβούλιο θα πρέπει να παρουσιάσει με διαφορετικό τρόπο κάποιες προτεραιότητες, οι οποίες θεωρεί ότι δεν είναι και τόσο προτεραιότητες, γιατί με τέτοιο πάγωμα εσόδων είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Η Αΐντα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα όλο το πρωί συζητούμε για τις πολιτικές που θέλουμε να υλοποιήσουμε τα επόμενα χρόνια. Μιλήσαμε για τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου, ποιε θα έπρεπε να είναι οι προτεραιότητες. Αλλά τώρα, αφού καθορίσαμε αυτά τα θέματα, θα πρέπει να δούμε πόσα κονδύλια θα δώσουμε για κάθε πολιτική και από πού θα τα βρούμε αυτά τα χρήματα. Αυτό το οποίο μπορεί κανείς να συνάγει ως συμπέρασμα από το κείμενο και τις τροπολογίες, μπορώ να πω ότι υπάρχει μεγάλη συνένεση ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτείται η πολιτική συνοχή επίσης και πολιτική όπως έρευνα, ανάπτυξη, ενέργεια, ενέργεια νεολαία, μεταφορές στα πλαίσια των στρατηγικών στόχων του 2020 θα πρέπει να έχουμε περισσότερα κονδύλια. Βεβαίως θα πρέπει όλες αυτές οι πολιτικές να χρηματοδοτούνται και από τις εθνικές προπολογισμούς και θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των προπολογισμών. Αλλά δεν θα πρέπει να αυταπατώμεθα, θα πρέπει να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση αυτών των πολιτικών και ο κοινοτικό προπολογισμό. Εξάλλου, στα πλαίσια στρατηγική 2020, και αυτό είναι κάτι το οποίο είδαμε σε όλε τι συζητήσει που είχαμε, είναι προφανέ το εξή. Δεν μπορούμε να επιβραδύνουμε το ρυθμό ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε να σταματήσουμε τι επενδύσει που είναι στρατηγική σημασία, ούτε τα διάφορα σχέδια που αφορούν το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουμε σημείο αναφορά παγκοσμίω. Διότι υπάρχουν άλλοι που μα περιμένουν στη γωνία. Η Ινδία, η Βραζιλία και η Κίνα. Και θα τρέξουν πιο γρήγορα από εμά. Θα πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου, αλλά θα πρέπει αυτή τη φορά η στρατηγική της Ευρώπης 2020 να τιμήσει τις θεσμεύσεις της, όχι να μας συμβεί ότι μας συνέβη με την στρατηγική της Λισαβόνης. Εμείς σε μια τροπολογία είπαμε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τις απαραίτητες πιστώσεις στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Βέβαια, λαμβάνοντας πάντα κατά νου το γεγονός ότι έχουμε περιορισμένες πιστώσεις στα πλαίσια του 1,29 των ΑΕΠ. Τώρα, τι σύστημα χρηματοδότησης και πού θα βρούμε αυτά τα κονδύλια για να χρηματοδοτήσουμε αυτό το 1,29 είναι κάτι που αποτέλεσε αντικείμενο τροπολογίας. Και λέμε ότι θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα ιδίων πόρων πραγματικό που σταδιακά θα υποκαταστήσει το παρόν σύστημα, στο οποίο αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό θα είναι η τέταρτη πίσω, δηλαδή ε, συνεισφορές των κρατών μελών που θα είναι ε, το ποσοστό αυτό του ΑΕΠ. Και θέλουμε με τον τρόπο αυτό να σταματήσουμε με την λανθασμένη και επιζήμια συζήτηση για τους που συνεισφέρουν ε, θετικά και αυτούς που συμφέρουν αρνητικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μελέτη αντικτύπων θα πρέπει να αφορά πού θα βρούμε αυτές τις νέες, ε, αυτούς τους νέους πόρους. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς, το έχουμε πει, θα πρέπει να γνωρίζουμε ε, τι θα γίνει στα πλαίσια αυτής της μελέτης και με το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ξέρουμε ότι είναι μία από τις καλύτερες εναλλακτικέ ε, λύσεις τις οποίες μπορούμε να υιοθετήσουμε. Πρώτα απ' όλα διότι σημαίνει ότι ο χρηματοπιστωτικός ε, τομέας θα πληρώσει ε, κατά κάποιο τρόπο για την κρίση που δημιούργησε. Επίση θα έχουμε πάρα πολλά χρήματα με αυτόν τον τρόπο, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο εφόσον γίνονται αυτές οι συναλλαγές αυτόματα να παίρνουμε το σχετικό ποσοστό. Σήμερα σε μια εφημερίδα λέει ότι χίλιοι οι οικονομολόγοι με μία επιστολή ζητούν από το G20 να το θέσει εφαρμογή. Καλύτερα να γίνει κατά την άποψή μας λοιπόν κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν λοιπόν κάνουμε αυτό το βήμα προς τα μπρος ως Κοινοβούλιο και ως Ευρωπαϊκή γενικότερα πιστεύω ότι θα μας ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες χώρες. Αυτές ε, είναι οι τροπολογίες που κατέθεσε η Σοσιαλιστική Ομάδα για το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ζητεί άλλο το λόγο. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε με τον εισηγητή ότι καταρχήν τα έσοδα θα πρέπει να στηρίζονται με συνέπεια στους ίδιους πόρους, ούτως ώστε να μην χρειάζονται πια ε, συνεισφορές από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αν συμφωνήσουμε και το γράψουμε και στο, στην έκθεση, θαυμάσια, να γίνει έτσι. Σαλβαντόρ. Πρόεδρε, σε σχέση με το μέγεθος του προϋπολογισμού, στην έκθεση αυτό το οποίο ζητούμε είναι το ανώτατο όριο για το 2013 να είναι το κατώτερο όριο για το 2014. Είναι μια θέση στην οποία θα αντισταθεί πάρα πολύ το Συμβούλιο που επηρεάζει πολύ τα πράγματα και ζητάει σε ονομαστική αξία πάγωνα. Άρα σε πραγματική αξία μείωση του προϋπολογισμού για τα επόμενα χρόνια. Εμείς δεν μπορούμε να, κάνουμε να πάμε σε διαπραγμάτευση με μια τέτοια πρόταση. Γι' αυτό εγώ στην έκθεσή μου ζητώ αύξηση 1,11% του κοινοτικού ΑΕΠ για τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Αυτό θα πρέπει να, θα πρέπει να είναι η βάση και οι υπόλοιπες ομάδες αναφέρονται αρκετά στο παρόν ανώτατο όριο των ίδιων πόρων, 1,23%. Και προφανώς αυτό είναι θεωρητικά το ανώτατο όριο, το πλαφόν στο οποίο μπορούμε να φτάσουμε. Τη στιγμή όμως που θα αρχίσουμε διαπραγμάτευση, ξέρουμε ότι θα πρέπει να φτάσουμε βάζοντας στο τραπέζι ένα εκατοστιαίο ποσοστό και με το 1,11 ξέρω ότι θα υπάρξουν συνάδελφοι και πολιτικές ομάδες που θα ζητήσουν κατώτερο ε, εκατοστιαίο ποσοστό, αλλά εγώ θέλω να αρχίσω με αυτό. Όσον αφορά τους ιδίους πόρους. Ξέρετε ποια είναι η θέση μου. Θα πρέπει να τιμήσουμε τις υποχρεώσεις και την εντολή που μας έδωσε η συνθήκη της Λισαβόνας, δηλαδή είμαστε μεταξύ των επιθυμιών και της πραγματικότητας, πιο κοντά στις επιθυμίες παρά στις πραγματικότητες θα έλεγα, δεδομένου ότι ακόμη είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο η όλη συζήτηση και τα κράτη-μέλη πρέπει να πω ότι πρακτικά δεν έχουν αρχίσει να συζητούν το θέμα αυτό. Ξέρετε ότι οποιαδήποτε απόφαση για την ε, μεταβολή των τρεχόντων ιδίων πόρων θα συνοδεύεται από τροποποίηση απόφασης για τους ιδίους πόρους, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινοβουλευτική επικύρωση από τους 27 διότι θέλουμε ομοφωνία, πράγμα που κάνει πολύ δυσχερή αυτή την όλη διαδικασία για νέους πόρους. Απ' την άλλη όμως υπάρχει γενική συνένεση στο Κοινοβούλιο και στην ΣΟΥΡΕ ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και να συζητήσουμε το θέμα των ίδιων πόρων. Υπάρχει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα αναλύσει πιο λεπτομεριακά την πρόταση αυτή και πιστεύω ότι εμείς ως πολιτική δήλωση λέγοντας ότι θέλουμε ιδίους πόρους και να μην υπάρχει το παρόν σύστημα το διορθωτικού προϋπολογισμού και των αντικαταβολών στα κράτη-μέλη, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Υπάρχουν τρία-τέσσερα υποχρεωτικά νούμερα τα οποία νομίζω ότι την χάνουν τις ε, συνένεσης των συναδέλφων του Κοινοβουλίου για τον κοινοτικό προπολογισμό. Η συμβιβαστική πρόταση λοιπόν η δική μου θα είναι πιο θεωρητική αν θέλετε από ό,τι πρακτική, αλλά διότι δεν έχω ε, συνένεση με Έχω επιτύχει συνένεση για συγκεκριμένο αριθμό. Θα πρέπει να συμφωνήσω την αρχή, με τη θεωρία. Και βεβαίω μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση με πραγματικούς αριθμούς για τις δαπάνε με το Συμβούλιο, αλλά για θέματα εσόδο σήμερα είμαστε στα χέρια του Συμβουλίου. Αν δεν θέλουν εκείνοι να ανοίξουν το όλο θέμα, μπορούμε να το επιτύχουμε με πλειοψηφία 500 στην Ολομέλεια, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες που έχουμε για το 2014 στον κοινοτικό προπολογισμό να μιλήσουμε για νέα έσοδα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση, για τις συνεισφορές των συναδέλφων και φεξής και μέχρι την επόμενη συνάντηση θα, θα προετοιμάσω με την γραμματεία ε, τις ε, Ήδη έχασα το πλάνο των 12, άρα μπορώ να αρχίσω από τώρα να δουλεύω θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες και οι συντονιστές επίσης θα δουλέψουν ταχύτερα. Τώρα για τις συζητήσεις με το Συμβούλιο για ενδεχόμενη αλλαγή του συστήματος ιδίων πόρων. Και εδώ εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξη. Ακούσαμε τη δήλωση της Κομισιόν που λέει ότι εν πάση περιπτώσει όταν ε, υποβάλει την νομοθετική της πρόταση τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου, ότι θα υποβάλει σχετικές προτάσεις για τροποποίηση του συστήματος ιδίων πόρων και το αργότερο τότε θα είναι η στιγμή που οπωσδήποτε πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα το Συμβούλιο και όταν διαπραγματευτούμε τις δημοσιονομικές προοπτικές ε, ως κοινοβούλιο, όχι ως σούρε, ως κοινοβούλιο, τότε θα πρέπει να μιλήσει το Συμβούλιο μαζί μας και για τους ιδίους πόρους. Έτσι νομίζω εγώ. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Και για πολλές ομάδες ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε την Μεγάλη Επανάσταση, την 1η Πρώτου του 2014, αλλά θα μπούμε σε μια εξελικτική διαδικασία. Αυτό μπορούμε να το θέσουμε ως στόχο μας. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άλλα πράγματα να συζητήσουμε, θα κάνω μερικές ανακοινώσεις. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθαν. Ε, προβαλόταν στο διαδίκτυο η συνεδρίαση από την Επιτροπή Γεωργίας, την Επιτροπή Γυναικών και την Επιτροπή Πολιτισμού ελάβαμε το μεταξύ τις γνωμοδοτήσεις τους. Εν μεταξύ είμαστε και πήγαμε σε κάποιες επιτροπές και ο Σαλβαντόρ και εγώ. Αυτή τη βδομάδα πήγα στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών και στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας. Η επόμενη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας θα λάβει χώρα στις 9 Μαΐου, όπου θα έχουμε μόνο μια μισή ώρα δουλειά και με πολύ συγκεντρωμένο τρόπο θα μιλήσουμε για την διοίκηση. Αυτό νομίζω ότι είναι επίσης πολύ σημαντικό και να ενημερώσετε όλους παρακαλώ. Δεν θα συζητήσουμε τίποτε άλλο πέρα από τη διοίκηση. Μια μισή ώρα στο Στρασβούργο. Δεν είναι πολύ το χρονικό διάστημα, αλλά για τη διοίκηση πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση οπωσδήποτε. Ελπίζω ότι ο εισηγητής θα κινηθεί αρκετά γρήγορα για να υποβάλει τις πρώτες προτάσεις του επί της συγχώνευσης κάποιων τροπολογιών και επί των συμβιβαστικών ενδεχομένως ώστε οι συντονιστές και οι σκιώδεις την επόμενη βδομάδα να μπορέσουν να συζητήσουν τα θέματα με τις ομάδες τους. Ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε και μείνατε μέχρι το τέλος και σας εύχομαι καλή ξεκούραση το Σαββατοκύριακο.